So, uh, dear, dear colleagues, ladies. Ε, ευχαριστώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Όρθιοι μόνο για χειροκροτήματα παρακαλώ, αλλιώς καθίστε. Uh, well, if I may open our hearing. Very important hearing. Energy costs and EU. Λοιπόν, έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ακρόαση. Το κόστος της ενέργειας και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ε, σας παρακαλώ, εκεί πέρα ο σύμβουλος των Πρασίνων, καθίστε. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντική η ακρόαση, όπως είπα. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Επίτροπο. Και σας ευχαριστώ για τις συζητήσεις. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Επίτροπο, τον κύριο Κανιέτε. Τα είπαμε και χτες και σήμερα το πρωί και στη συνάντηση με τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες και σας ευχαριστώ όλους εξ ονόματος Επιτροπής που δεχτήκατε να έρθετε σε αυτήν την ακρόαση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως οι ανακατατάξεις των τιμών είναι πάρα πολύ σοβαρές, ειδικά του πετρελαίου που είχε πάει σε πολύ ψηλά επίπεδα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα είναι τόσο χαμηλές που δεν καλύπτεται το κόστος της εξόριξης ε, σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι τα στοιχεία των αγορών. Βεβαίως η προσφορά και η ζήτηση που επηρεάζουν, αλλά και άλλα. Ως συνήθως ε, σε μια ελεύθερη αγορά, τα μεταφορικά, η ασφάλεια, αλλά και κάποια στοιχεία της πολιτικής. Όπως οι επιδοτήσεις, ε, φορολογία κτλ. Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ακρόαση για να δούμε ποιο είναι το κόστος ε, της ενέργειας και το πώς επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα. Προβλέπονται 2,5 ώρες, θα έχουμε δύο τμήματα στη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε τις εταιρίες ε, και την οικονομική διάσταση και το άλλο αφορά τους χρήστες της ενέργειας. Οι δραστηριότητες μας λοιπόν ε, δεν γίνεται να αφορούν μόνο τους ε, καταναλωτές και να μην περιλαμβάνουν τις εταιρείες. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ζητήσω από τους ε, ειδικού μας ε, και τους ε, βουλευτές μας να είναι σύντομοι γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να ζητήσω από τον κύριο Κανιέτη, τον Επίτροπο, να κάνει κάποιες πρώτες παρατηρήσεις πριν περάσουμε στην ακρόαση. Κύριε Επίτροπε, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι χαρά μου που ξαναήρθα ήρθα τόσο σύντομα αυτή τη φορά να μιλήσουμε για τις ε, τιμές της ενέργειας και το πώς επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι σημαντική πολιτική ανησυχία, επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και επηρεάζουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα. Όπως ξέρετε, η Επιτροπή μας είχε ένα σαφή στόχο να ξεκινήσει ξανά να αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή οικονομία. Βεβαίω συστάθηκε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για να έχουν οι επιχειρήσεις πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Βελτιώνουμε επίσης ε, την ε, ένωση των ε, χρηματαγορών και ρίχνουμε τα διάφορα εμπόδια και φραγμούς που υπάρχουν. Αλλά το κόστος της ενέργειας παραμένει ένας τομέας που έχει πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα. Και είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρώπη ακόμα δεν έχει κάποιο πλέον έκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές μας. Η Ενεργειακή Ένωση θα μας βοηθήσει να φτάσουμε εκεί και βέβαια η στρατηγική είναι να χρησιμοποιήσουμε την μετάβαση της ενέργειας για να σταματήσει η εξάρτησή μας από τα ορεικτά καύσιμα. Μέχρι να συμβεί αυτό πάντα θα είμαστε ευάλωτοι στις παγκόσμιες αγορές ε, και την κινητικότητα των τιμών. Τα καλά νέα είναι πως πλησιάζουμε στον στόχο μας. Είμαστε πρώτοι στον κόσμο σε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν αποδοτικά την ενέργεια. Και άρα ο σχετικό κλάδος αυτή τη στιγμή απασχολεί γύρω στα 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές ε, οικολογικού σχεδιασμού υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσουν 100.000 επιπλέον θέσεις εργασίας και 54 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020 και οι εταιρείε μα ε, από τις καλύτερες στον κόσμο παίζουν σημαντικό ρόλο στις εταιρείε, στις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας. Το κόστος των ηλιακών πάνελ έχει μειωθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά μας. Υπάρχει λοιπόν πρόοδος, αλλά γεγονό είναι πως αυτή η μετάβαση δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, οπότε πρέπει να δούμε το πού βρισκόμαστε σήμερα. Και αυτό σημαίνει να αντιληφθούμε πως ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές τιμές της ενέργειας και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική και επίκαιρη αυτή η ακρόαση και γι' αυτό η Κομισιόν προετοιμάζει αυτή τη στιγμή μια συνέχεια στην έκθεση του 2014 για το ενεργειακό κόστος. Πριν αναφερθώ στο τι μπορούμε να αναμένουμε στη φετινή έκθεση, θα ήθελα να ξαναδώ τα βασικά ευρήματα του 2014 και να εξηγήσω πώς η Ενεργειακή Ένωση αναφέρεται σε αυτά. Τα ευρήματα της έκθεσης του 2014 ήταν εντυπωσιακά. Ήταν πως το κενό η ψαλίδα μεταξύ των τιμών στα διάφορα κράτη μεγάλωνε. Οι καταναλωτές σε κάποια κράτη-μέλη πλέον από 2,5 έως 4 φορές περισσότερο από άλλα κράτη-μέλη. Και σε κάποιες περιπτώσεις οι τιμές ε, βενζίνης και ηλεκτρισμού ήταν πολλαπλάσιες ε, των ΙΠΑ και βλέπουμε πως οι τιμές λιανικής ε, του ηλεκτρισμού αυξάνονται κατά 3,5% το χρόνο και για φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό οι τιμές λιανικής ε, αυξάνονταν και αυξάνονταν και το κομμάτι τους που ήταν φόροι και τέλη. Και μάλιστα σε χώλες με υψηλή διείσδυση ηλιακής ε, και αιωλικής ενέργειας υπήρχε μία μείωση των τιμών ενώ σε άλλες όχι. Θα πρέπει λοιπόν τη μέση χοντρική να συγκλίνουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προτείναμε αυτό. Δεν συνέβη όμως στην ε, τιμή της ε, λιανικής. Γιατί έχουμε τους ε, φόρους, τα τέλη, τους διαφορετικούς κανονισμούς, τους διαχειριστές του δικτύου που διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Με τις προκλήσεις αυτέ. η συστάση μας ήταν σαφής. Χάρη στην Ενεργειακή Ένωση ήδη κάνουμε σημαντική πρόοδο. Δείτε φέτος. Το πακέτο για την ε, ασφάλεια της ε, παροχής ε, εστιάζεται στο να γίνει η αγορά του φυσικού αερίου πιο προβλέψιμη και ανταγωνιστική. Πέρσι μόλις εστιαστήκαμε στο να αρχίσουμε να οικοδομούμε τις υποδομές που χρειάζεται η αγορά μας για να κρατήσουμε χαμηλές τις τιμές. Έτσι θα βελτιωθεί η διαχείριση του δικτύου και θα υπάρχει καλύτερη διασύνδεση λιανικών και χονδρικών αγορών. Επίσης εξετάζουμε την τιμολόγηση του άνθρακα μέσω του σχεδίου για το εμπόριο εκπομπών και την μεταρρύθμισή του και βέβαια θα καλύψουμε τους τομείς που δεν καλύπτονται ήδη από αυτό. Θα προτείνουμε μια ενημέρωση της ε, σχετικής οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικές και όσον αφορά το κόστος ενέργειας εστιάζουμε στο να μειώσουμε την κατανάλωση και την ζήτηση. Γι' αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να περάσουμε νομοθεσία για την αποτελεσματική χρήση της ενέργειας. Θα πρέπει λοιπόν να μειωθούν οι τιμές και να μας βοηθήσουν και οι εταιρείες να διαχειριστούμε το κόστος ενέργειας. Θα πρέπει να βελτιωθεί η αξιοπιστία, η αηφορία και η προβλεψιμότητα της παροχής ενέργειας για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Όλα αυτά βεβαίως είναι σημεία πρόοδου, αλλά το οποίο άλλαξε πάρα πολύ έκτοτε. Γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε στη φετινή έκθεση θα Βλέπουμε πως η τιμή του πετρελαίου πέφτει και το ίδιο βεβαίως ε, και η τιμή του ηλεκτρισμού. Η τιμή των ορεικτών καυσίμων έχει μειωθεί κατά το 1 τρίτο και οι τιμές της είναι μόνο διπλάσιες ε, από τις ΙΠΑ και βλέπουμε πως οι τιμές ε, των ορεικτών καυσίμων Όσον αφορά τις εισαγωγές, μειώθηκαν από 400 δισεκατομμύρια ευρώ το 2013 σε 260 δισεκατομμύρια το 2015. Μία μείωση 35% σε δύο χρόνια. Η μείωση των εισαγωγών μεταξύ 2013 και 2014 κατά 140 δισεκατομμύρια ισοδυναμεί με 1% του ΑΕΠ της Ένωσης. Βεβαίω ε, το ότι το ευρώ εξασθένησε γιατί η ισοτιμία του έπεσε από 1,40 το Μάιο 2014 σε 1,06 το 2015 ήταν τη τάξη του 24% σε 10 μήνες και άρα αυτό αντιστάθμισε κάπως ε, την ε, μείωση της τιμής των ορεικτών καυσίμων. Βεβαίω. Κάποια από αυτά οφείλονται και στην ε, πολιτική μας, καθώς αυξήθηκε η αποτελεσματικότητα και οι τεχνολογίες για να μειωθεί το κόστος και κάποια σχετίζονται με εξωτερικούς παράγοντες. Το σχιστολιθικό αέριο των ΙΠΑ μπήκε στην αγορά, έχουμε δυναμική ανάπτυξη στην Ασία και νέες χώρες που εμφανίζονται στην αγορά. Τέλος πάντων οι τιμές αυτές μας δίνουν κάποιο περιθώριο στο μακροοικονομικό επίπεδο και δίνουν στην βιομηχανία μας, ιδιαίτερα την ενεργοβόρα βιομηχανία, την ευκαιρία να επενδύσει σε νέες τεχνολογίες. Όμως θα ήθελα να είμαι σαφής. Αυτό το οποίο δεν κάνουν αυτές οι τιμές είναι να μας ε, δώσουν την ευκαιρία να χαλαρώσουμε. Γιατί το μόνο σίγουρο είναι πως οι τιμές αυτές δεν θα παραμείνουν εκεί που είναι. Παραδείγματος χάρη, οι τιμές σήμερα είναι περίπου αυτές που ήταν το 2009 και το 2012 ήταν γύρω στο 120 δολάρια το βαρέλι μεταξύ 2004 και 2008 ανέβηκε από τη σημερινή τιμή στα 140 δολάρια το βαρέλι. Τι εννοώ. Ε, οι τιμές αλλάζουν γρήγορα γι' αυτό ως συνέχεια της έκθεσης του 2014 δεσμευτήκαμε να ξεκινήσουμε μια τακτική παρακολούθηση των τιμών της ενέργειας. Η έκθεσή μας για το 2016 θα δημοσιευτεί το καλοκαίρι και θα δει τις τάσεις των τιμών, τις διεθνείς ρυθμίσεις, αλλά και το τι γίνεται μεταξύ κρατών μελών. Θα καλύπτει και τα νοικοκυριά και τη βιομηχανία, αλλά και τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Θα θέλαμε λοιπόν να ακούσουμε στο δυνατόν περισσότερες πήγες ε, και ενδιαφερόμενους. Ακούσαμε τον Ιανουάριο, είχα μια τέτοια πρώτη συνάντηση, διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και τώρα θέλουμε να ακούσουμε και εσάς. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στόχος αυτών των αναλύσεων είναι να είμαστε στο δυνατόν πιο ενήμεροι για να προετοιμάσουμε μια κατάλληλη αντίδραση και να έχουμε μια σαφή εικόνα του αντικτύπου στην ε, αηφορία της Ευρώπης. Οπωσδήποτε η έκθεση αυτή θα μας βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη της κατάστασης και να δούμε την πρόοδο που την Αναμένω να ακούσω τις απόψεις σας και να συνεργαστούμε στις πρωτοβουλίες που έρχονται για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Mr. Commissioner. Uh, Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ξέρουμε ότι ο Επίτροπος έχει χρόνο μέχρι τις 4. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε γρήγορα. Θέλουμε να ακούσουμε τις εμπειρογνώμονές μας, καταρχήν, και εν συνεχεία θα γίνουν ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο κύριος Μπασκουνιάν είναι ο πρώτος ομιλητής. Τι περίπλοκο ισπανικό όνομα είναι αυτό. Γενικά τα ισπανικά ονόματα. Αλλά μάλλον, καλά το είπα, ε. ο οποίος ε, έκανε σπουδέ οικονομικών, αλλά πριν από έξι χρόνια εξελέγει ε, δικη, ε, διευθυντής μιας εταιρείας και αντιπρόεδρος της ε, European Wind Association και είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής ε, Υπηρεσίας ε, Αιωλικής Ανέργειας τα τελευταία δύο χρόνια. Ενδιαφέροντα τα όσα έχετε κάνει. Είσαστε υπεύθυνο για τις ανανεώσιμες λοιπόν και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Είναι προνόμιο που εκπροσωπείται η Αξιώνα σε αυτή τη δημόσια κρόαση. Η σημερινή συζήτηση είναι πολύ σημαντική και είναι σημαντική γιατί η συζήτηση για το αν η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης τίθεται να αμφιβόλει λόγω του κόστου της ενέργειας ξεπερνάει μια συζήτηση για τη βιομηχανία της Ευρώπης. Ορισμένοι λένε ότι η πολιτική για το, για το κλίμα και την ενέργεια θα πρέπει να μειώσει τις φιλοδοξίες λόγω της αρνητικής επιπτωσής στην ανταγωνιστικότητα. Εμείς ε, τα μελετήσαμε αυτά και θα έχουμε και ένα νέο έγγραφο σύντομα από την Κομισιόν. Γι' αυτό δεν σκοπεύω να βασιστώ στα τελευταία δεδομένα και δεν μπορώ να πω και ποια είναι η τελική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Απλώ θα πρέπει να μιλήσω για κάποια θέματα που πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε. Ε, είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία αυτή που εκπροσωπώ που ασχολείται με τι ανανεώσιμε ενέργειε. Από αυτή τη σκοπιά θα μιλήσω. Για να βελτιώσουμε την οικονομία και την ε, ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη είναι να ε, εντατικοποιήσουμε τις πολιτικές μας για ένα νέο ε, ενεργειακό ε, πλαίσιο για τις μας. Δύο λόγια για την εταιρεία μου, την Ακθιώνα. παράγουμε 8,5 ΜΒ σε όλο τον κόσμο, σε 20 χώρες, 7 ευρωπαϊκές και είμαστε η πέμπτη εταιρεία παραγωγής ολικής ενέργειας πέραν των ε, Κινέζων. Όλα αυτά ξεκίνησαν πριν λίγα χρόνια. Ε, θεωρούμε ότι είμαστε ένα καλό παράδειγμα του πώς η ευρωπαϊκή πολιτική ανανεώσεων βοηθάει τις ευρωπαϊκές εταιρείε και τη βιομηχανία να δώσει νέα προϊόντα και να γίνουν παγκόσμιοι παίκτες. Να πάω στο συγκεκριμένο θέμα, το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν δύο διαφορετικοί ορισμοί τη ανταγωνιστικότητα. Πρώτον, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, είναι οι θεσμοί, οι πολιτικέ και οι πτυχέ που καθορίζουν το επίπεδο ε, ευημερία σε μια χώρα. Αυτό ε, εξαρτάται από πολλά πράγματα. Ε, χρηματοπιστωτική ικανότητα, σταθερότητα κτλ. Απ' την άλλη, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα είναι κάτι πολύ πιο περιορισμένο. Ε, είναι η ικανότητα μια δεδομένη βιομηχανικού κλάδου να ανταγωνιστεί. Αυτό επηρεάζεται από πολλούς ε, διαφορετικούς ε, παράγοντες, ε, το κόστος των κρατικών χεριών, φορολογία, το κόστος των πρώτων υλών κτλ. Και το κόστος ενέργειας είναι ένα από αυτά τα στοιχεία που επηρεάζουν όμως την ανταγωνιστικότητα μιας εταιρείας. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι πρέπει να χωρίσουμε την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας μιας βιομηχανίας από το θέμα της γενικής ανταγωνιστικότητας. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και το θέμα δούμε ποιοι κλάδοι ε, έχουν, πληρώνουν πολύ για την ενέργεια. Ε, το ΑΕΠ, αυτές οι, αυτές οι, αυτοί κλάδοι ε, συνεισφέρουν στο 1,4 του συνολικού ΑΕΠ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι πολύ σημαντικό. Ε, οι βιομηχανίες οι οποίες είναι δάσος ενέργειας γενικά ε, περιορίζονται. Και είναι λογικό επίσης γιατί η Ευρώπη δεν έχει ενεργειακούς πόρους. Πέρα από τις ανανεώσιμες βέβαια. Το δεύτερο μήνυμα είναι λοιπόν ότι η ανταγωνιστικότητα των κάποιων βιομηχανικών κλάδων δεν αφορούν την συνολική βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Οι βιομηχανίες που δαπανούν πολλή ενέργεια σίγουρα και το πόσο ανταγωνιστικέ είναι είναι τεράστιο θέμα για την Ευρώπη, αλλά δεν αφορά ολόκληρη τη βιομηχανία τη Ευρώπη, όλου του κλάδου τη Ευρώπη. Αφού εντοπίσουμε του ε, βιομηχανικού τομεί όπου χρειάζεται να εστιάσουμε, πρέπει να καθορίσουμε ποιο είναι το κόστο τη ενέργεια. Και εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κόστος τη ενέργεια έχει δύο διαφορετικέ συνιστώσει: το κόστο για το φυσικό αέριο και το κόστο για, για το ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρική ενέργεια. Και το μερίδιο του φυσικού αερίου στην ε, παραγωγή ενέργειας είναι ψηλότερο από τις ε, ηλεκτρικής ενέργειες Αυτό φαίνεται από διάφορες μελέτες. Του 2014, ας πούμε, τη μελέτη της Κομισιόν μέχρι ε, την ε, πρόσφατη μελέτη που έγινε από μια εταιρεία consultant για τις 25 πρώτες εταιρείες. Και το φυσικό αέριο ε, έχει μεγαλύτερο μερίδιο στο κόστος της ενέργειας. Ε, επίσης υπάρχει η εξέλιξη του σχιστολιθικού αερίου, του μεριδίου που έχει το σχιστολιθικό αέριο στην, α, της Αμερικής. Την προσοχή μας συνήθως τη δίνουμε στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα όμως στο φυσικό αέριο, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε σωστά το πρόβλημα όταν αποφασίζουμε τις επιλογές της πολιτικής μας. Σωστό είναι ότι όμως δεν θα πρέπει να λησμονούμε και τα προβλήματα της, του ηλεκτρικού ρεύματος. το ηλεκτρικό ρεύμα α, γίνεται όλο και πιο ακριβό τελευταία. Παρότι γενικά ήταν πιο σταθερό, ειδικά για μεγάλους ε, βιομηχανικούς καταναλωτές από το 2012 με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Επομένως, το θέμα είναι σε ποιο βαθμό αυτό το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζει αυτούς τους βιομηχανικούς τομείς και την ανταγωνιστικότητά τους, που είναι πολύ ενεργοβόροι. Για να απαντήσουμε, ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε διάφορα πράγματα. Καταρχάς, οι ενεργοβόρες εταιρείε πληρώνουν πολύ λιγότερα από τα νοικοκυριά ή τους μέσους ε, βιομηχανικούς καταναλωτές για την κατανάλωσή του. τα νοικοκυριά πληρώνουν για την ηλεκτρική ενέργεια δύο, μισή φορές παραπάνω από τις ενεργοβόρες εταιρείε και οι μικρές βιομηχανικέ εταιρείε πλέον 40% ε, παραπάνω. Ε, επίσης, οι τιμές τη της ενέργεια ενέργειας για τις ενεργοβόρες εταιρείε διαφέρουν πάρα πολύ από κλάδο σε κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι λοιπόν, υπάρχει ένα και μόνο πρόβλημα ή έχουμε πολλαπλά προβλήματα με διαφορετικά κόστη. Τρίτον, όπως βλέπετε από, από την, το μπλε οι ενεργοβόρες εταιρείε ε, πληρώνουν για το λεκτικό ρεύμα ε, τιμές που καθορίζονται από την αγορά. Και αυτό συνδέεται με τις, τιμές, τις αγορές τιμές και πολύ λιγότερο με τους φόρους και τα τέλη. Όπως είπε και η Κομισιόν, και ο Επίτροπος μάλλον, ε, το κόστος των εργατικών χεριών και το κόστος των φόρων και των δασμών καθορίζονται πολύ από τις ε, πολιτικές επιλογές. Οι ενεργοβόρες ε, εταιρείες και καταναλωτές εξαιρούνται από το κόστος αυτό σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή. Αυτοί οι τομεί ε, υποφελούνται δηλαδή σε πολλέ χώρε από τη μισιακή μεταχείριση σε ό,τι αφορά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο. Επιπλέον, ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλα εργαλεία όπω ε, δωρεάν ε, ποσοστώσει, α πούμε, και πολλά άλλα εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί και τις έχει, τα έχει λάβει υπόψη τις μελέτες της Κομισιόν. Το τέταρτο μήνυμα είναι λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να εξετάσουμε όλα αυτά προσεκτικά όταν μελετάμε αν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα ε, ανταγωνιστικότητας για αυτούς τους κλάδους ε, στην Ευρώπη και ποιο είναι ο λόγος για αυτό το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας ε, λόγω του κόστους. Ε, και αν συνδέονται με τη στρατηγική του κλίματος και της ενέργειας της Ευρώπης και τις σχετικές πολιτικές. Επίσης, μην ξεχνάμε ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής, που είναι η πολιτική για τις ανανεώσιμες ενέργειες σε αυτούς τους ε, βιομηχανικούς τομείς. Μερικές φορές οι ανανεώσιμες πηγές θεωρούνται ανταγωνιστικές προς την, ε, και αντίθετες με την τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Δεν είναι σωστό. Το έγγραφο εργασία Κομισιόν 2014 λέει, ε, μας δείχνει κάποια ανησυχητικά πράγματα ε, για δύο τομεί, ε, όπως το χλώριο και το αλουμίνιο. 0,9 και 2% ήταν το κόστο ε, της ενέργειας. Αυτό δεν φαίνεται να είναι τρομερό ποσοστό. Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε την επίπτωση των ε, κάποιων επιπτώσεων που μετριάζουν το κόστος. Παραδείγματο χάρη η σημασία της ε, αιωλική ενέργειας και της ε, αιωλική ενέργειας που όταν μπαίνουν στην αγορά μειώνουν τις τιμές γενικά της ενέργεια, ε, όσο πιο πολύ διδίνουν οι ανανεώσιμε, τόσο πολύ μειώνονται οι τιμές. Και όσο ψηλή είναι η συμμετοχή τους στο τιμολόγιο, τόσο πιο λίγα πληρώνουμε. Αυτό μπορεί να έχει θετική επίπτωση σε στενοκοβόρες βιομηχανίες όπως ε, δείχνει στη σελίδα 9 η ανακοίνωση της Κομισιόν του 2014. Η επί... το καθαρό, η καθαρή επίπτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ότι, όπω φαίνεται στην Ισπανία και στην Ιρλανδία, μειώνουν τελικά τι τιμέ και δεν τι αυξάνουν. Βλέπετε τη ε, σχέση ανάμεσα ε, στο επίπεδο διείσδυσης των ανανεώσιμων και στο επίπεδο των τιμών της ενέργειας. Όσο περισσότερο διδεί η αιωλική ενέργεια στην ισπανική αγορά, και αυτά είναι τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2014, τόσο πιο χαμηλή η τελική τιμή. Και πιο χαμηλό το τιμολόγιο για τον ενεργοβόρο καταναλωτή. Δύο λόγια τώρα για την αρχή της παρουσίασης μου. Τι γίνεται με την ε, γενική ανταγωνιστικότητα. Για μας που ασχολούμαστε με τις ανανεώσιμες, που δεν υπήρχαν πριν από 20 χρόνια, είναι σαφές ότι η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εταιριών ε, στην Ευρώπη βοηθά την οικονομία και θα το κάνει ακόμα περισσότερο εάν ε, υλοποιήσουμε τους στόχους του μέχρι το 2030. Επομένως, αν υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, θα πρέπει να λυθεί σωστά. Και αν οι πολιτικοί αποφασίσουν να βρουν κάποιο, κάποια λύση στο πρόβλημα, θα πρέπει να το κάνουν μετά από ανάλυση και να ληφθούν υπόψη οι υπόλοιπε ε, ενεργειακές και κλιματικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε για τα πάρα πολύ σαφή μηνύματα που αν τα αρρύθμισα σωστά ήταν πέντε. Για να δούμε και τα δικά σας πέντε σημεία των υπολείπων. Σας ευχαριστούμε ε, σας και πάμε στον δεύτερο, τον καθηγητά, καθηγητή κύριο Κάρστεν Νόιχοφ, φυσική, στο Πανεπιστήμιο της Εδελβέργης, LSE, Cambridge και καθηγητής ενέργειας και κλιματική αλλαγής στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Πολυτεχνείο του Βερολίν. Υγείται πολλών project ε, για τις ε, αλλαγές του κλίματος και διεξάγει μελέτες σε πολλούς τομείς ε, και για το ETS μεταξύ άλλων. question is very, very important. Είναι πολύ σημαντικό ε, αυτά που λέω. Οικονομική διάσταση, πάροχη ενέργειας. Για πείτε μας εσείς και από την εμπειρία σας. Αλλά μην ξεπεράσετε και τα 10 λεπτά σας παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με προσκαλέσετε. Και τα δικά μου 5 cent. Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των όσων παράγουν υλικά και άλλων βιομηχανικών φορέων. Δεύτερον, η εξέλιξη των τιμών των καυσίμων και των πρώτων υλών. Το είπε και ε, ο Επίτροπος. Πρέπει να έχουμε ανταγωνιστικότητα και εδώ στην πολιτική μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ρευστότητα των τιμών, να χρησιμοποιήσουμε τις ανανεώσιμες επειδή είναι χαμηλή η τιμή των ορυκτών καυσίμων σήμερα, μεγάλη ευκαιρία για την Ευρώπη και τρίτον, πρέπει να δούμε και να εφαρμόσουμε στην πράξη το δυναμικό καινοτομίας και αποτελεσματικότητας. Πάντα με φόντο την μείωση των τιμών πετελαίου. Βλέπετε εδώ μια εικόνα που χαρακτηρίζει το μερίδιο του ΑΕΠ στην περίπτωση της Γερμανίας σε σχέση με το μερίδιο του συνολικού κόστους. Και τι σχέση έχει το κόστος ενέργειας με αυτό το συνολικό είναι 10, 20 και 30 στον κάθετο άξονα. Και στον οριζόντιο βλέπετε 2% περίπου του ΑΕΠ της Γερμανίας και δεξιά κάτω στον ε, κάθετο, στον οριζόντα άξονα γύρω στο 1,6 κατά μέσο είναι το ποσοστό και διάφορα ε, υλικά έχουμε εδώ, χάλιβας, βασικά χημικά, αλουμίνιο κτλ. Μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες. Και έτσι μπορούμε να εστιάσουμε σε αυτά τα υλικά και νομίζω ότι αυτή είναι μια νέα συζήτηση γιατί πάντα κάναμε μια διάκριση σε ό,τι αφορά την ένταση της ενέργειας αλλά νομίζω πιο εύκολο είναι με τις ύλες, με τα υλικά. Εδώ βλέπετε τα βασικά, αυτά είναι τα σημαντικά. Αν δείτε στην υπόλοιπη βιομηχανία, είναι πιο σημαντική για την Ευρώπη, αλλά για, την, για τον υπόλοιπο κλάδο, τους υπόλοιπους κλάδους ε, της βιομηχανίας 98% ε, του ΑΕΠ. Το ενεργειακό κόστος δεν είναι στρατηγικό, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε τις επόμενες αυτούς κλάδους για να βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοσια. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ήθελα να ε, αναφέρω διάφορα το προετοίμαζα την ομιλία μου. Κυρίως, επαναλαμβάνω, πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις χαμηλές τιμές ε, στο πετρέλαιο ιδίω, αλλά και στο φυσικό αέριο. Είναι δραματική μείωση των τιμών του πετρέλαιου και του φυσικού αερίου, ε, ιδίως στο, στην περίπτωση του πετρελαίου. Μειώνεται και η παγκόσμια ζήτηση. Έχει σχέση ε, μέρη όλο το φαινόμενο αυτό και με την ενεργειακή απόδοση. Πάντως το αποτέλεσμα είναι σχετικά μικρή συνιστόσα σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Επίσης βλέπαμε τριπλάσεις από τη ΣΥΠΑ, πολύ ψηλές πάντως τιμές για το φυσικό αέριο και εδώ πάλι να έχουμε μείωση. Ε, η μικρή απόλυτη διαφορά πλέον σε σχέση με το φυσικό αέριο. Άρα εκεί που διαφοροποιεί το πάρα πολύ η κατάσταση στην Ευρώπη ε, βλέπουμε να μην υπάρχει διαφορά. Και για τον άνθρακα έχουμε μείωση γιατί έχουμε πλεονασματική παραγωγή και έχουμε τις τιμές ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Αν επιβάλλεις ε, μία τιμή πάνω στο διοξίδιο βλέπεις ότι ε, μειώνεται και η τιμή του άνθρακα. Τώρα, να συζητήσουμε το κόστος της πολιτικής ό,τι αφορά το κόστο των υλικών, είναι σχεδόν ανύπαρκτο αυτό. Αν δούμε τις τιμές τώρα της ισχύω. Εδώ είναι πιο μεγάλη η διακύμανση. Ανατολική ακτή, είπα, είναι η πράσινη γραμμή και οι άλλες γραμμές είναι διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Πώς θα αντιμετωπίσει ο κλάδος αυτή τη ρευστότητα, αυτή τη διακυμάνσεις. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάποιες δυνατότητες hedging, κάλυψης, αντιστάθμισης. Μπορεί να υπάρχει αυτή η διακύμανση σε κάποιους κλάδους της βιομηχανίας σε ένα δεδομένο έτος, σε κάποιους άλλους, σε κάποιο άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και με τους πληστριασμούς, ε, να έχουμε κάποιες συμβάσεις ε, hedging, είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτό. Και επίσης, βλέπετε εδώ τις ε, εναλλαγές των τιμών μέσα στην ίδια μέρα. Πιστεύουμε στο μέλλον θα προσλάβει μεγαλύτερη σημασία αυτή η συνιστόσα. Και για τις ενεργοβόρες βιομηχανίας μέρος της παραγωγής θα μπορούσε να μετατοπιστεί στις περιόδους που είναι χαμηλότερη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Και άρα μειώνουμε και το μέσο όρο της τιμής του ηλεκτρισμού. Βέβαια πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρώτη της αλλά και άλλα στοιχεία. Πρέπει να είμαστε καινοτόμοι και να προχωρήσουμε. Αλλά με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι βελτιώνουμε την ενεργειακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Ανανεώσουμε πηγές ενέργειας. Σε αυτό το διάγραμμα κάτω-κάτω βλέπετε με το μπλε τι έχουμε δαπανίσει ε, με το, ε, για τις εισαγωγές καυσίμων ορυκτών με το κόκκινο το εγχώριο και με τον γκρι βλέπετε τις εκπομπές δοξιδίου του άνθρακα. Βλέπετε να πέφτουν οι τιμές ε, το 2015. Ποια είναι τώρα η μαύρη αυτή η διάστηκτη γραμμή Εδώ έχουμε δύο τρίτα ε, ολική ενέργεια και ένα ηλιακή. Και είδαμε τις επενδύσεις. Δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε εύκολα, αν το ε, βλέπαμε στο παρελθόν, σε αυτή τη σύγκριση. Αλλά σήμερα φτάνουμε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, όπως βλέπετε. Και γι' αυτό είμαι και αισιόδοξο για την ασφάλεια της ενέργειας, για την πολιτική, για το κλίμα και για τις θέσει εργασία, Γιατί μπορούμε όλα όσα εξάγουμε να τα δαπανίσουμε αυτά τα χρήματα για να ε, προωθήσουμε τις επενδύσεις στην Ευρώπη σε αυτούς τους τομείς ενέργειας που σας ανέφερα. Ας υποθέσουμε όμως, ο υπολογισμός έγινε με βάση την υπόθεση ότι το σταθμισμένο κόστος του κεφαλαίου ήταν 5%. όταν πήγαμε σε Ευρωπαίους επενδυτέ και του είπαμε το 2014 ποιο είναι το σταθμισμένο κόστο για, για την ολική ενέργεια και σχετικά project, βλέπετε στην ε, Γερμανία ήταν 3,5 με 4,5%, σε αλλε ηταν ήταν 8-9%, στην Ελλάδα ήταν 12%, αλλά και σε χώρε όπως τη Σουηδία ήταν 8%. Ποιε είναι οι επιπτώσει, Για να πάμε στην προηγούμενη εικόνα. Αν δεν έχουμε αυτό το 5% αλλά έχουμε 4% σταθμισμένο κόστος όπως στη Γερμανία ε, αυξάνουμε το κόστος της ε, απαλλαγής από τον άνθρακα δεν επιτρέψουμε την κάλυψη και την αντιστάθμιση με διάφορα συμβόλαια ειδικά και άμα φτάσουμε όπως στη Σουηδία που είναι 8 στο 10-12% τι θα γίνει με την απαλλαγή ε, από τον άνθρακα. Γίνεται πιο δαπανηρή αυτή η πολιτική. Άρα ποιε είναι οι επιπτώσεις στην Ευρώπη. Θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να υπάρξει συνεργασία. Όσε δηλαδή χώρε έχουν υψηλότερο κεφαλαιακό κόστο να βοηθηθούν ώστε να μειώσουν αυτό το κόστο. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε και με την ΕΤΕΠ και με κοινά project. Τέλο πάντων, να εκμεταλλευτούμε τι επενδυτικέ ευκαιρίε σε αυτέ τι χώρε. Θα πρέπει να εστιάσουμε στο σχεδιασμό πολιτικής για τη δημιουργία ενός ε, καλού επενδυτικού πλαισίου. Υπάρχουν πολιτικές ε, που μπορούν να βοηθήσουν, όπως η πολιτική των ε, αμοιβών. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν πολύ δαπανηρές, τώρα είναι πιο φθηνές. Πρέπει να κάνουμε το σχετικό υπολογισμό, πρέπει να έχουμε αυτή την αμοιβή, αυτή την ανταμοιβή για τις ανανεώσιμες πηγές, για να μειώσουμε το κόστος. Επίσης, αποφασίσαμε, μάλλον ε, σχεδιάσαμε και συζητήσαμε τι ανανεώσιμε θεωρώντα ότι είναι πάρα πολύ δαπανηρέ, ώστε πάντα θα απαιτείται στήριξη. Βλέπετε όμω τι διακυμάνσεις, Είδαμε και στο προηγούμενο γράφημα. Πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι θα αυξηθούν οι τιμέ στο μέλλον. Ε, των ορυκτών καυσίμων. Μπορεί να παραμένουν χαμηλέ για ένα-δύο χρόνια. Αυτέ είναι εκτιμήσει, αλλά θα σταθεροποιηθούν και μάλλον θα σημειώσουν αύξηση στα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα είδο ασφάλεια, εξασφάλιση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε του καταναλωτέ, γιατί είναι μια αμφίδρομη συμφωνία μεταξύ των χρηστών ενέργεια και των ανανεώσιμων. Ε, τώρα έχουμε κάλυψη τι χαμηλέ τιμέ ε, ε, των καυσίμων και πρέπει μετά να προστατεύσουμε του καταναλωτέ από την αύξηση αυτών των τιμών. Τώρα, τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ ευραίων κλάδων τη βιομηχανία, το 1,6 με το συνολικού κόστου είναι το ενεργειακό κόστο, αλλά να δούμε και άλλε πτυχέ. Και θέλουμε πρότυπα που θα βοηθήσουν για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίε και δυνατότητε. Γι' αυτό και έχουμε στόχου, έχουμε διαδικασίε στην Ευρώπη. Πάμε στον τομέα των υλικών, όπου το ενδιακό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ειδικέ διατάξεις και είναι πολύ ελπιδοφόρα αυτή η προσέγγιση. Να περάσουμε σε ένα σύστημα benchmark ε, σε ό,τι αφορά το ETS και την αντιστάθμιση της τιμής ε, της ισχύω. Βέβαια μιλάμε μόνο για την παραγωγή και για διαδικασίε που βελτιώνουν την απόδοση. Τι βλέπουμε τώρα, εξυγχρονισμό, μετριασμό. Έχουμε ε, σε αυτέ τι διαδικασίε ε, αξία, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι τα εργαλεία μετά το Παρίσι που θα ε, προωθήσουμε και με το ETS και σε ό,τι αφορά εξαιρέσει στον τομέα αυτό. Και έρχομαι στο τελευταίο σημείο. Για να εκμεταλλευτούμε τις επαναστατικές τεχνολογίες, το ETS δεν θα μας βοηθήσει θα πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε τέτοιες επαναστατικές τεχνολογίες. Θα πρέπει να επενδύσουμε. Έχουμε τα ταμεία, ταμεία συγχρονισμού, αλλά θα πρέπει να υπάρξουν κοινέ στρατηγικές της βιομηχανίας και των κυβερνήσεων. Γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο τομέας των υλικών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Διαφοροποίηση λοιπόν μεταξύ του τομέα των υλικών και άλλων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ε, η ανάπτυξη των τιμών της ενέργειας που μας δίνει αυτή τη στιγμή ευκαιρία που δεν πρέπει να τη χάσουμε. Θα πρέπει να βοηθήσουμε επίσης ε, τη βιομηχανία να αντισταθμίσει αυτή, αυτές τις διακοιμάσεις, τις δύο σε ευκαιρία. Θα πρέπει να φροντίσουμε επίσης να τα μπορούσουμε να περάσουμε ε, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά με χαμηλό κεφαλαίο κόστος και επίσης θα πρέπει να έχουμε και ειδικά προγράμματα για το μίσο όπως είναι ο άνθρακας και τα υλικά και για τους άλλους γενικότερα να έχουμε άλλε άλλες διατάξεις για το γενικότερο τομέα της ενέργειας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω πως μετράτε και πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Τα έχω σημειώσει όλα. Τώρα ήρθε η ώρα για ερωτήσεις και απαντήσεις. Λοιπόν, ο κύριος Πίπερ, πρώτα απ' όλα από το ΕΛΚ. If I may ask you, uh, I ask you maybe two minutes questions, all of us, because we don't have too much time. Δύο λεπτά ο καθένας, γιατί δεν υπάρχει χρόνος δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την λεπτομερέστατη ενημέρωση όσον αφορά το κόστος. Κοιτάξτε, κάποια πράγματα μου ξέφυγαν, γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νόιερ. Όταν έχουμε μέσες επιχειρήσεις, μέσες βιομηχανίες, ιδιώτες ε, στον ηλεκτρισμού. Ε, ε, δεν μπορούμε τώρα δηλαδή να εμπιστευτούμε κανένα στατιστικό στοιχείο. Νόμιζα ότι παγκοσμίω ε, η Ευρώπη είναι στην κορυφή. Προσπαθήσατε να μας πείτε πως ε, δεν είναι τόσο άσχημη η κατάσταση και πως οι τιμές σε παγκόσμια σύγκριση δεν είναι τόσο κακές που να εμποδίζουν τον ανταγωνισμό. Η δεύτερη ερώτησή μου αναφέρατε την ενεργειακή αποδοτικότητα για να περιορίσουμε την εξάρτηση. Ναι. Βεβαίω ε, το θέμα είναι ότι αυτά τα υπολογίζεται με μια επέκταση των ΑΠΕ, αλλά έχουμε κάθε χρόνο υποχρέωση για εξοικονόμηση κατά 1,5% και για τις ΑΠΕ. Μήπως με αυτές τις πολιτικές ε, προκλήσεις μας εμποδίζουμε την καλύτερη και αποδοτικότερη ανάπτυξη των ΑΠΕ. γιατί υπάρχει μια γενική υποχρέωση εξοικονόμησης ε, και για τις ΑΠΕ. Και μας είπατε μετά, εντάξει δεν είναι τόσο χάλια τα πράγματα κτλ. Εγώ ακριβώς αυτό θεωρώ το κόστος της ε, πολιτικής, ε, δηλαδή κάνουμε τη ζωή μας δύσκολη. και υπάρχει μη αποδοτικότητα. Εγώ λοιπόν είδα πολλές αντιφάσεις στην παρουσίασή σας και θα ήθελα να μας ε, τα εξηγήσετε αυτά. Ευχαριστώ, Νταν Νίκα, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και θα ήθελα να τον ρωτήσω ε, αν μπορεί να μας εξηγήσει λίγο τις ε, δηλώσεις ε, που έγιναν. Ο κύριος Λόπες είπε πως δεν υπάρχει πρόβλημα με την ανταγωνιστικότητα. Μετά είδαμε ότι η τιμή της ενέργειας της ΕΠΑ είναι η μισή από αυτή που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, θεωρώ πως δεν είναι πάρα πολύ χρήσιμο να διατηρηθεί μια κατάσταση η οποία δεν επηρεάζει την πραγματικότητα, γιατί Όλα αυτά δίνουν πάτημα σε όσους θέλουν να σκοτώσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Το βασικό στοιχείο που επηρεάζει τις ε, ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές, είναι το ότι υπάρχει ένα πλαφόν στον κλάδο. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως πρέπει και υπάρχει μια διατάραξη των τιμών συνέργειας, προφανώς οι ανανεώσιμες ε, πηγές ε, ενέργειας ε, δεν θα προωθηθούν. Δηλαδή πώς θα φτάσουμε το στόχο του 20% όταν δεν συζητάμε καν τις τιμές για αυτούς που θα πρέπει να έχουν ένα σύστημα εφεδρικό. Θεωρείτε ότι μπορούμε να φτάσουμε 100% ΑΠΕ και θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό είναι ψέμα, γιατί ακόμα και η Κομισιόν λέει ότι αν θέλουμε να ξεπεράσουμε το 30% χρειάζονται ε, κάποιες ε, ειδικέ συνθήκες. Και βεβαίω ε, τη στιγμή που δεν φυσάει ο αέρας ή δεν λάμπει ο ήλιος θα πρέπει να έχουμε ενέργεια. Λοιπόν, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια έχουν ένα σύστημα με βάση το οποίο λειτουργούν, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να στραφούμε σε άλλε πηγέ. Ή να κλείσουμε τα συμβατικά εργοστάσια παραγωγή για να στραφούμε σε ΑΠΕ. Πρέπει να τα λάβετε υπόψη αυτά. Ο πρόεδρο διακόπτη, σα ευχαριστώ, κύριο Χένκελ από το Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση. Ο πρώτο μιλητή είπε πως οι ανανεώσιμες δεν επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών. αυτό ισχύει γιατί πληρώνει κάποιος άλλος. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος πληρώνει. Στη χώρα μου φαίνεται πως ε, για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, χάνουν ανταγωνιστικότητα. Και τα νοικοκυριά επίσης ε, στη χώρα μου συνεισφέρουν γιατί οι τιμές της ενέργειας ηλιανική δηλαδή για τα νοικοκυριά είναι η δεύτερη υψηλότερη στην Ευρώπη στη Γερμανία. Θα ήθελα λοιπόν ξεκάθαρα να σας ρωτήσω ποιος πληρώνει έτσι ώστε οι ενεργοβόρες βιομηχανίες να μην υποφέρουν από το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ευχαριστώ κυρία Πόνσερ, νέα βουλευτής ε, των φιλελευθέρων στην Επιτροπή μας. Καλώς ήρθατε. Κυρία μου, έχετε το λόγο. Για τον κύριο Κανιέτη είναι η ερώτησή μου. Μια άμεση ερώτηση. Μιλήσατε για το κόστος της, των ανανεώσιμων. Των ανανεώσιμων. Ε, και όχι, θέλω να ξέρω, εάν έχει, έχετε υπολογίσει το πόσο μειώνουν το, τις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη οι ανανεώσιμες πηγές όταν διεισδύουν. Και επίσης και ποιο είναι το, το κόστος των ανανεώσιμων, όχι μόνο η μείωση. Από τους πράσινους. έγινε μια μελέτη για τις γερμανικές ενεργοβόρες ε, βιομηχανίες και το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Βλέπετε απάνω την ε, χονδρική αγορά που επωφελείται από τις ανανεώσιμες κατά 10 ευρώ, δηλαδή ε, οι ανανεώσιμες κάνουν την ανανεώσιμη οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κάνουν την χονδρική αγορά πιο φθηνή στη Γερμανία στο μέσο βλέπουμε την αντιστάθμιση για τις έμεσες επιπτώσεις του ETS που αντισταθμίζεται από τα έσοδα από τη δημοπρασία. Ε, το κόκκινο είναι η φόρη και το μπλε είναι το κόστος του δικτύου που κανονικά πληρώνουν οι καταναλωτές στη Γερμανία αλλά η γερμανική βιομηχανία ε, έχει 80% μεγαλύτερη μείωση από τους υπόλοιπους. Και το αποτέλεσμα αυτής της μελέτης δείχνει ότι οι γερμανικές ενεργοβόρες βιομηχανίες πληρώνουν σήμερα, φυσικά εξαρτάται από την τιμή χοντρικής, κάτι μεταξύ 32 και λιγότερο από 32, εάν μειωθούν τιμές χοντρικής. Επομένως, το γεγονός ότι οι ανεώσιμες μειώνουν το κόστος ισχύει πέρα από τη Γερμανία και στην Ισπανία και πώς το εξηγείτε. Και κυρία Νόεχοφ. εσείς ως Γερμανός πιστεύετε ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι σωστά. Θέλω περισσότερες λεπτομέρειες για τις τρεις ιδέες σας. Τι μπορούμε να κάνουμε για τις ενεργοβόρες ε, εταιρείε, για το hedging, δηλαδή για την αντιστάθμιση κινδύνου. Ποιος θα αναπτύσσει αυτά τα προγράμματα. Επίση θα πρέπει να βασιστούμε, να λάβουμε υπόψη μα μάλλον, ε, τι τιμέ και το κόστο του κεφαλαίου. Κύριε Νίκα, μιλήσατε για ένα ταμείο που συνδέεται με το ταμείο του Γιούνκερ, που θα εξασφαλίσει το, θα καλύψει το κεφαλαιακό κόστο ε, στη Νότια Ευρώπη. Γιατί, αν ας πούμε πληρώσετε ε, για την αιωλική ενέργεια ε, το κόστος του κεφαλαίου για την επένδυση δηλαδή είναι 4% ενώ αν θες να επενδύσεις στη Γερμανία, στην ε, Ρουμανία ας πούμε το κόστος του κεφαλαίου, δηλαδή το κόστος της επένδυσης είναι 8%. Μακάρι να ήταν κάποιοι από τους εργάτες της Χαλιβουργίας ε, εδώ ε, να ακούγαν τη συζήτηση γιατί απολύθηκαν. Και ένας λόγος που κλείχαν οι εταιρείε είναι ότι είχαν ψηλό κόστο, είχε ψηλό κόστος η ενέργεια περίπλοκος σύνδεσμος επιδοτήσεων, ε, στόχων, ε, ποσοστώσεων κτλ. σημαίνει ότι είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε την τιμολόγηση. Διερωτώ αν οι τιμές που αναφέρεται για τις ανανεώσιμες είναι το άμεσο κόστος ε, από την αιωλική κτλ. Ή έχετε συμπεριλάβει το κόστος για την ανάπτυξη δυναμικού, τις αλλαγές του δικτύου και όλα τα άλλα μεγάλα κόστη που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε τις διαλύψατες που έχει το δίκτυο. Κλείνεται όμως ε, αξιόπιστα εργοστάσια που παράγουν ενέργεια με σταθερό ρυθμό και τα αντικαθιστάτε με εργοστάσια που παράγουν έτσι απρόβλεπτες ποσότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για μιλήστε σας παρακαλώ με τα βιομηχανίες χημικών, αλουμινίου, χάλιβα κτλ που τι κάνουν, κλείνουν τα εργοστάσια στην Ευρώπη, ε, μετακινούνται εκτός Ευρώπης. Ε. Έχουμε ένα νέο πρόγραμμα αλλαγή του συστήματος εμπορίας εκπομπών που σχεδιάζεται ειδικά για να αυξήσει την πίεση σε αυτούς τους operator. Γνωρίζετε εσείς ε, ομιλητές ότι η επίπτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι όχι να μειώσει τις εκπομπές, αλλά απλώς να εξάγει τις εκπομπές και συχνά τις εξάγει σε άλλες χώρες με χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα, όπου οι εκπομπές αναμονάδα παραγωγής είναι υψηλότερες και έχουμε τελικά μια πολιτική η οποία υποσκάπτει την ευρωπαϊκή οικονομία και αυξάνει τις ε, παγκόσμιες εκπομπές. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι έξυπνη πολιτική. Ευχαριστώ. Η κυρία Λόπες Μπερμέρο από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Αναμφίβολα η τιμή της ενέργειας είναι ουσιώδες ζήτημα για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Το ίδιο ισχύει και για τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ανταγωνισμό από άλλες χώρες με χαμηλότερο εργασιακό περιβαλλοντικό κοινωνικό κόστος. Γι' αυτό και η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να εμπαθύνουμε σε αυτό με νέες εμπορικές συμφωνίες. Δράτω με τις ευκαιρίες για να ρωτήσω τους ε, ομιλητές, ιδίως για το σε κρίση όπως είναι η Χαλιβουργία για παράδειγμα, σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι η παραγωγή, η διανομή κτλ. στην αγορά ηλεκτρισμού θα μπορούσε να ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε χωρίς να απαρνηθούμε τους στόχους ενεργειακής απόδοσης και της πρόθεση ανανεώσιμων πηγών να μην προκαλέσει ε, επιπλέον κόστος για τους καταναλωτές στη χώρα μου. Την Ισπανία, για παράδειγμα, ε, δεν υπάρχουν βιομηχανικά τιμολόγια ε, και είναι πολύ μεγάλη η τιμή της ενέργειας σε σχέση με τη μέση τιμή του, του ρεύματος για τα νοικοκυριά. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μετακυλήσουμε το κόστος στους καταναλωτές από τις τεχνολογικές προσαρμογές που είναι αναγκαίες για πιο καθαρές τεχνολογίες. Θα πρέπει να έχουμε δημόσιες πολιτικές μεταξύ άλλων που θα φρενάρουν την δύναμη του ολιγοπολίου στο τομέα του ηλεκτρισμού. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό το πρόβλημα υπάρχει μόνο στην ε, χώρα μου ή σε άλλες ή στην Ευρώπη εν γέννη και αν ξέρετε καλές πρακτικές ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρισμού που θα διατηρεί τη βιωσιμότητα του κλάδου και θα μπορεί αυτός να συμβάλλει στο ευρωπαϊκό παραγωγικό μοντέλο μέσω ε, τιμολογίων προσαρμοσμένων ή μέσω άλλων μεθόδων παραγωγής προσαρμοσμένων σε ανάγκες. Ευχαριστώ. Κυρία Πιλάρ Καστίγιο, ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε ουσιαστικά για το κόστος της ενέργειας. Και στο πλαίσιο μιας πραγματικότητας που ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη για την εσωτερική αγορά ενέργειας μιλάω. Είναι ένα άλλο στοιχείο. Ένας παράγοντας που δεν θα πρέπει να παραλείψουμε σε αυτή τη συζήτηση. Από αυτήν την έννοια είναι αναπόδραστο να συζητήσουμε ένα θέμα που έχει διάφορες οπτικές γωνίες και δυνατότητες. Για παράδειγμα, μηχανισμοί αντιστάθμισης. Διαφορετικές φόρμουλες και τύποι ό,τι αφορά αυτούς τους μηχανισμούς αντιστάθμισης που δημιουργούν κάποιες συνθήκες ανταγωνισμού που δεν είναι ίδιες πάντα. Θα ήθελα λοιπόν ο Επίτροπος, οι εισηγητές να μου πούν πώς βλέπουν την ανάγκη ή όχι να φτάσουμε όχι απαραίτητο σε εναρμόνιση, αλλά τέλος πάντων σε έναν μεγαλύτερο συντονισμό αυτών των θαυμιστικών μηχανισμών. Θεωρείτε ότι είναι κάτι απαραίτητο ή δεν έχει τόση σημασία για, τη, για τον προσδιορισμό του κόστους. Thank you very much, madam. Ε, Ευχαριστώ. Ο κύριος Έριξον. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσες ήταν οι παρουσιάσεις. Πρέπει να μας συγχωρήσετε μας τους πολιτικούς. Γιατί όταν εκλεγόμαστε λέμε ότι η Ευρώπη φταίει που είναι τόσο ψηλές οι τιμέ τα κτλ. Και μετά που έχουμε εκλεγεί βλέπουμε ότι υπάρχουν άλλα πράγματα. Και τελικά δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι εύκολο και να προσαρμοστούμε στην αλλαγή της πραγματικότητας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κανιέτε, δεν θα πολύ καλό τα συμπεράσματα αυτά, επί παραδείγματι, να προωθήσουμε περισσότερο αιωλική ενέργεια μες γενιένη ή προγράμματα για εισαγωγή των ανέσμων με χαμηλότερο κεφαλαιακό κόστος. Δεν θα ήταν, επαναλαμβάνω, πολύ καλό να έρθετε σε επαφή με αυτές τις χώρες που σήμερα έχουν πολύ, μεγάλη, πολύ ψηλά τιμολόγια για τον ηλεκτρισμό και την ενέργεια εν γέννη, Πολωνία, Πορτογαλία, Ενωμένο Βασίλειο. Δεν θα έπρεπε να τις πιέσετε να θετήσουν στρατηγία μείωση του κόστους. Να προσθέσω κι εγώ μια ερώτηση προς τον κύριο Λόπες. Είπατε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του κόστους ε, του φυσικού αερίου και του κόστου πετρελαίου. Πολύ απλά σας θέτω το εξής ερώτημα. Αυτό που οφείλεται την πρωτογενή ενεργειακή πηγή, το φυσικό αέριο και με την, ε, ενώ με τον, από τον ηλεκτρισμό μπορούμε, τον ηλεκτρισμό να τον παραγάγουμε από διάφορες πηγές όπως ουράνιο, ορυκτά, καύσιμα, ενάνωσες πηγές ενέργειας, ένας φορέας ενέργειας, δηλαδή ηλεκτρισμός. Αυτή, αυτός είναι ο λόγος της τόσο μεγάλης διαφοράς του κόστους, εν γέννη, στην περίπτωση φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Επίτροπε, να θέσω και σε εσά ε, αυτά τα ερωτήματα ε, και θα ήθελα να ακούσω και τις παρατηρήσεις σας. Θα σας δώσω πρώτα το λόγο σε εσά επειδή ξέρω ότι θα πρέπει να φύγετε. Ας ε, προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κόστος της ε, ενέργειας ε, μέσα στην Ευρώπη, πώς επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα, τι γίνεται με τη απέ αν είναι παράγοντας που αυξάνει ή μειώνει την ανταγωνιστικότητα. Και έχουμε ανακατέψει δύο διαφορετικές συζητήσεις, πώς θα αναπτύξουμε τις ΑΠΕ και ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά το ενεργειακό κόστος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Οι τιμές ε, της ενέργειας ε, παγκοσμίω είναι υψηλότερες από αυτές των ανταγωνιστών μας. Είναι σαφές πως υπάρχουν κάποιες βιομηχανίες που χρησιμοποιούν περισσότερη ενέργεια, κάποιοι μίλησαν για τα υλικά και ανέφερε τους κλάδους, ε, κάποιοι είναι ενεργοβόροι, άλλοι λιγότερο ενεργοβόροι. Στο σύνολο όμως της Ένωσης, εάν συγκρίνουμε το τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο και τις τιμές του στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιανουάριο του 2016. Στο NBP του Ηνωμένου Βασιλείου η τιμή ήταν δύο φορές ψηλότερη από το αντίστοιχο τέρμιναλ στη ΣΥΠΑ. Πριν από τρία χρόνια ήταν τριπλάσια και τετραπλάσια. Τώρα είναι μόνο η διπλή. Αλλά βεβαίω είναι πάλι πρόβλημα ότι είναι διπλάσια. Και πρέπει να το λύσουμε. 2012 ήταν 3,5 φορές παραπάνω. Στο αέριο λοιπόν έχουμε... Μικρότερο πρόβλημα. Στον ηλεκτρισμό. Πριν από λίγα χρόνια είχαμε μια αναλογία 2,5 με 3,5 ε, φορές υψηλότερες τιμές από ό,τι στη ΣΥΠΑ. Τα τελευταία τρίμηνα του 2015 ήταν στο 1,6. Οπότε υπήρχε τεράστια ψαλίδα, έχει μειωθεί. Υπάρχει όμως ακόμα ψαλίδα. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός της αγοράς ηλεκτρισμού, οπωσδήποτε και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός ε, στην αγορά αερίου με μια στρατηγική LNG, με διαφορετικές διαδρομές, με διασυνδέσεις για να μειωθεί η ψαλίδα. Υπήρχε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Κάποιος ρώτησε το τι, πώς επηρεάζουν η ΑΠΕ την τιμή και την βιομηχανία. Αν δείτε το τι συμβαίνει με την τιμή του ηλεκτρισμού στη βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τιμή για τον βιομηχανικό καταναλωτή από το 2014 μέχρι 2018 αυξήθηκε κατά 11%. Οι τιμές αυξάνονται λοιπόν. Το 2015 η αύξηση ήταν ε, λιγότερη. Αλλά εάν αναλύσουμε πού οφείλεται η αύξηση της τιμής, φόροι και τέλη είναι το 66% της αύξησης. Τέλη δικτύου 23%. Και το κομμάτι της ενέργειας μειώθηκε κατά 4%. Α, κάτι πιο κομμάτι μπορεί να έχει σχέση με τη ΣΑΠΕ, αλλά δεν έχω αυτή τη λεπτομέρεια αλλά δεν είναι οι ανανεώσιμες που μπαίνουν στο σύστημα αυτές οι οποίες φταίνε για την αύξηση της ε, τιμής. Δεν είναι η ΑΠΕ, είναι άλλα στοιχεία. Γιατί έχουμε ένα περίπλοκο σύστημα. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή, ότι έχουμε το διπλάσιο κόστος από τους ανταγωνιστές μας και πρέπει να αναπτύξουμε τις ΑΠΕ και να γίνει αγορά κατάλληλη για ΑΠΕ γιατί η αγορά μας και η αγορά που έχουμε είναι σχεδιασμένη για κεντρική παραγωγή με ορυκτά καύσιμα από λίγες εταιρείες. Τώρα θα έχουμε πολλούς παραγωγούς με αποκεντρωμένη παραγωγή με ανανεώσιμες. Είναι διαφορετική η κατάσταση και χρειάζεται διαφορετική αγορά. Οπότε το πιο δύσκολο νομοθέτημα φέτος ε, στην Επιτροπή σας θα είναι ο σχεδιασμός αγοράς για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και μετά υπήρχε το ζήτημα του εάν το σύστημα εμπορίας εκπομπών είναι υπεύθυνο για την κρίση ε, στο χαλιβουργία. Μα ας είμαστε σοβαροί, το πρόβλημα της χαλιβουργίας δεν είναι τα 5 ευρώ τον τόνο η τιμή του άνθρακα, είναι ο ανταγωνισμός από την Κίνα, η υπερβολική δυναμικότητα, 300 εκατομμύρια τόνου, 300 εκατομμύρια τόνοι υπερβάλλουσα παραγωγή στην Κίνα και η Κίνα θα λάβει και το καθεστώς οικονομίας της αγοράς και γνωρίζει η Κομισιόν ότι πρέπει να προστατεύσουμε τη βιομηχανία μας αλλά υπάρχουν οι κανόνες του ΠΟΕ. Το πρόβλημα για μένα είναι να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας. Αυτό είναι το βασικό. Και να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με τις μελέτες της Κομισιόν. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποια διαρροή ανθρακά λόγω, λόγω του συστήματος εμπορίας εκπομπών. Από άλλους παράγοντες ναι, αλλά όχι από αυτό το λόγο. Γιατί οι πιο εκτεθειμένη κλάδη έντασης ε, ενέργειας ε, θα έχουν ούτως ή άλλως ε, δωρεάν άδειε και θα καλύπτονται. Οι άλλοι κλάδοι θα έχουν μικρότερο επίπεδο προστασίας. Αυτή είναι η γενική εικόνα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή την έκθεση τελικά γιατί μπορούμε να αντλήσουμε διάφορα διδάγματα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να συζητήσουμε ακριβώς το κόστος της ενέργειας στην Επιτροπή μας που είναι αρμόδια για την ενέργεια. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τώρα. Να ζητήσω από τους ε, εμπειρογνώμονες μας να απαντήσουν τις ερωτήσεις μας. Αποφασίστε δημοκρατικά. Ποιο θέλει πρώτος να μιλήσει. Δημοκρατικά δίνω το λόγο στο Γερμανό ομιλητή. Αρχίζω από τα σχόλια του κύριου Πίπερ. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για τις τιμέ ενέργειας και την ανταγωνιστικότητα τη βιομηχανία, γι' αυτό ε, εστίασα στις ενεργοβόρες βιομηχανίε, που είναι σημαντικό στοιχείο οι τιμέ για την ανταγωνιστικότητα. Σε άλλους κλάδους βιομηχανία. αν έχουμε ενεργειακό κόστος 1,6% του τζίρου, αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό για την ανταγωνιστικότητα. Το ενεργειακό κόστο σίγουρα είναι σημαντικό για μικρέ επιχειρήσει και για τα νοικοκυριά βέβαια. Είδαμε λοιπόν την αλλαγή για τα νοικοκυριά στη Γερμανία, για παράδειγμα. Στη δεκαετία του 90 τα νοικοκυριά δαπανούσαν 2,2% το εισοδήματό του ε, για το ρεύμα. Τώρα ε, αυτό το ποσοστό έχει ανέλθει στο 2,5%. Υπήρξε αύξηση λοιπόν και οι απνανέσουμε πηγέ ενέργεια ευθύνονται, αλλά πάλι έχουν μια ισορροπία. Για τα φτωχά νοικοκυριά η πρόκληση είναι μεγαλύτερη, αλλά υπάρχουν μηχανισμοί για να αντιμετωπιστεί. Αυτό που πρέπει να κατανοήσετε είναι ότι η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία και σε κάποιο βαθμό και η Τσεχία επένδυαν ε, στα φωτοβολταϊκά και στην αιωλική ενέργεια ε, στην αριστερή πλευρά του γραφήματος όταν οι τεχνολογίες αυτές ήταν πολύ πιο δαπανηρές 40 σέντ ανά κιλοβατόρα για τις επενδύσεις σήμερα είναι 10 ή 8 σέντ και γι' αυτό έχουμε σε χώρες όπως η Ισπανία, η Γερμανία, αυτές τις, ε, αυτά, αυτά τα νούμερα. Δεν τη δημιουργήσαμε τις τεχνολογίες όταν ήταν ε, δαπανηρές, έχουμε μάθει όμως. Η επένδυση αυτή έγινε, θα έλεγα, από πολιτικό ατύχημα στις χώρες αυτές, αλλά τελικά σημείωσε παγκόσμια επιτυχία. Όποια χώρα αντιμετώπισε αυτή τη στρατηγική δεν θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, γιατί το κόστος της τεχνολογίας πλέον έχει μειωθεί. Για τον κύριο Νίκας, ναι, πράγματι, ήταν απλουστευμένη η εικόνα και ρητά και ξεκάθαρα είπα ότι εξαιρείται το συστημικό ενεργειακό κόστος ε, για τις δύο συνιστός. Αν έχουμε το σύστημα των ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να έχουμε επενδύσεις ε, στην παραγωγή, στο δίκτυο κτλ. Παρ' όλα αυτά, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η όλη συζήτηση ήταν η πρωτογενή ε, παραγωγή ενέργεια με ΑΠΕ. Ήταν πολύ δαπανή και αυτό έχει αλλάξει. Αν εχουμε 5 5-6% ΑΠΕ, Νομίζω ότι με αυτό το σενάριο θα πρέπει να ε, κάνουμε πιο ελαστικούς, ευέλικτους τους χρήστες της ενέργειας και να έχουμε ολοκλήρωση του συστήματος ενέργειας στην Ευρώπη. Είναι από πλευράς πολιτικής ε, μια προσπάθεια που απαιτεί ιδιαίτερη ένταση. Και όταν περνάμε από το 70-80% στο 100% ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, θα επενδύσουμε πολύ σε πεντρικέ δυνατότητε, για φυσικό αέριο, στην αποθήκευση, θα πρέπει να επενδύσουμε. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε υπόψη μα αυτό το ποσοστό 80% του περίπου για τι ΑΠΕ. Ένα άλλο ερώτημα ήταν ακριβώ για το hedging, για αυτή την αντιστάθμιση. Βλέπουμε στι σχετικέ συμβάσει στη Γερμανία για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ότι έχουμε αρκετά καλή ρευστότητα και διάρκεια αυτών των συμβάσεων, μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη, μικρή συμμετοχή ιδιωτικών φορέων στι γειτονικέ χώρε. Αν χρησιμοποιηθεί η τιμή αυτή για την ε, αντιστάθμιση, ο κίνδυνος στο ρίσκο είναι μεγαλύτερο. Άρα θα πρέπει να είναι της ίδιας διάρκειας ε, οι συμβάσεις ε, για να είναι δυνατή αυτή η αντιστάθμιση. Άρα θα πρέπει και σε πραγματικό χρόνο και στην ίδια ημέρα να έχουμε αυτή την πλήρη ισχύ μετάδοσης, μεταβίβασης. Από ευρωπαϊκής πλευράς λοιπόν τα συμφέροντα και εμπειρίες των αντιονταλικών χωρών ε, και ε, Πολωνία και Ελλάδα, Ιταλία <clears throat> είναι πολύ σημαντικές. Ενώ η εμπειρία στην ε, Δυτική Ευρώπη διαφέρει. Για τον κύριο Χέλμ. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στον κλάδο της Χαλιβουργίας και καταλαβαίνω την ερμηνεία σας ότι έχει μειωθεί από το 2008 κατά 20% η ζήτηση χάλιβα και δεν πρόκειται να ανακτήσει αυτό το χαμένο έδαφος ο τομέας. Έχουμε αυξημένες καθαρές εξαγωγές ε, χάλιβα όμως. Άρα κατάλαβαν τελικά ε, ότι έπρεπε να κλείσουν κάποιους, ε, κάποιες μονάδες. Έγινε αυτή η επιλογή. Τώρα αν προχωρήσουμε Έχουμε και την Κίνα. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με την Κίνα, να πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στον τομέα αυτό. Για τη διαρροή άθρακα. Αφού έχουμε αύξηση των καθαρών εισαγωγών, δεν έχουμε πρόβλημα με διαρροή άνθρακα. Το αντίθετο έχουμε. Για την κυρία Καστίγιο. η συνεργασία για τις εξαιρέσεις θα είναι κάτι σημαντικό. Και αυτή η προσέγγιση με το ETS και την αντιστάθμιση των τιμών είναι ένα σημαντικό επίσης Πρέπει να ορίσουμε κάποια κατώτατα όρια, κάποια benchmarks. Ένας τόνος χάλιβα ή ένας τόνος αλουμινίου είναι ένας τόνος. Ε, με τα υλικά δεν έχουμε πρόβλημα. Όμως, αποτύχαμε παταγωδός ε, στις ανανεώσιμες. Και ήταν στρατηγικό λάθος στην ΚΔ ανταγωνισμού τότε. Πήγε πάρα πολύ γρήγορα. Και ξανά άνοιξε πράγματα που ήταν εκτός των ορίων. Και μπήκαν και πολιτικά ζητήματα. Και τελικά υπήρχαν κάποιες οδηγίες για κρατικές ενισχύσεις και εξαιρέσεις. Και η Γερμανία έπρεπε να είναι τελικά πιο αστήρη με τι εξαιρέσει. Άρα εκεί δεν τα πήγαμε καλά, αποτύχαμε. Πρέπει να Υπάρξει λοιπόν μια πολιτική διαδικασία και δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. And now I would like to ask our... Our... Και τώρα. Ο κύριος Λόπες θα απαντήσει. Αξιώνω να το λέτε, Πρόεδρε. Είναι πολύ πιο σύντομο. Θα απαντήσω στις ερωτήσεις που μου απευθύνανε οι ευρωβουλευτές. Ο κύριος Νίκα λέει ότι οι ανανεώσιμες δεν επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα. Εγώ ε, είπα ότι την επηρεάζουν λιγότερο από, άλλοι από άλλους παράγοντες, ειδικά και τις ενεργοβόρες ε, βιομηχανίες. Και αν αυτό δεν το λάβουμε υπόψη στην ανάλυση, τότε οι αποφάσεις θα είναι λανθασμένες. Γιατί οι ανανεώσιμες ε, πηγές ενέργειας δεν ε, είναι υπεύθυνε για τα προβλήματα ανταγωνιστικότητα ε, τη Ευρώπη. Μπορείτε να τι ξεφορτωθείτε. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα είναι αναποτελεσματικό για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των ενεργοβόρων ε, επιχειρήσεων. Με το να επιτεθείτε στι ΑΠΕ δεν πρόκειται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων εταιριών. Μάλιστα, εγώ νομίζω ότι όσο πιο πολλέ ανανεώσιμε έχουμε στην αγορά, τόσο πιο χαμηλέ οι τιμέ. Αυτά λένε οι ειδικέ μελέτε και τη Κομισιόν. Κύριε Χίνκλου. Όπως και προλαλή σας. Εγώ εστίασα στην επίπτωση του κόστους ενέργειας στις ενεργοβόρες ε, ε, βιομηχανίες, γιατί είναι και πιο σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης γενικά. Δηλαδή, ουσιαστικά θέλησα να εστιάσω στο μεγάλο κομμάτι του προβλήματος. Πόσο πληρώνουμε για τις ανανεώσιμες τώρα. Σε πολλές ε, χώρες πληρώνουμε μηδέν. Γιατί το τα μακροοικονομικά νούμερα διαφόρων χωρών δείχνουν ότι θα πρέπει φυσικά να πληρώσεις ε, για την υποστήριξη προ τις ανανεώσιμε. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν, γιατί έχουν πολλά ωφέλη στην ενεργειακή σου αγορά, ε, στις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και στην οικονομία σου. Όσο μεγαλύτερη δίδυση των ΑΠΕ, μπορεί να έχει αυτά τα, τις θετικέ επιπτώσει. επιπτώσεις, όπως στην Ισπανία, όπου επηρεάσα, ε, λά, λάβαμε υπόψη τις τιμές των ε, ανανεώσιμων, των εισαγωγών, κάναμε τη σύγκριση και είδαμε ότι είναι θετική επίπτωση. Το θέμα είναι πόσο πληρώνουμε ακριβώς γι' αυτό. Είναι σαν να λέτε πόσο πληρώνετε για την οικοδόμηση δυναμικού. χρειαζόμαστε όλο αυτό το δυναμικό. Γιατί είμαστε υπέρ, χωρίς να ξέρουμε πόσο ακριβώς δυναμικό χρειαζόμαστε οι πληρωμέ που δίνουμε σε αυτές και τα ωφέλη που δίνουμε σε αυτέ τι εταιρείε είναι δίκαια και τι γίνεται με τον άνθρακα. Τι γίνεται με τι περιφερειακέ επιδοτήσει που, που περιλαμβάνονται στους, σε ενεργειακά τιμολόγια. Τι γίνεται με τι κοινωνικέ πολιτικέ, πόσο κοστίζουν. Πόσο δίκαιε είναι αυτέ οι πολιτικέ και άρα το κόστο του. Ε, το να πληρώνουμε για τι ΑΠΕ είναι πολύ πιο δίκαιο από το να πληρώνουμε για άλλα πράγματα. Γιατί τελικά όλοι μαζί πολεμάμε την καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής και την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, που ξέρουμε θα μας φέρει πολλά οικονομικά προβλήματα. Φυσικά, φυσικά μην ξεχνάμε και την ανταγωνιστικότητα, αλλά μην θεωρείτε τα υπόλοιπα δεδομένα. Έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλες πτυχές. δε Δικαστήριο. Για το συντονισμό. Είναι καλό, καλή ευκαιρία για να προωθήσουμε κάποιους μηχανισμούς συντονισμού. Το πρόβλημα με την ευρωπαϊκή αγορά είναι ότι δεν υπάρχει μία αγορά στην Ευρώπη. Αν υπάρχει πλήρη συντονισμό και ενοποίηση τη αγορά και αν το πιέσουμε αυτό το πράγμα, μπορεί να μην έχουμε καλά αποτελέσματα. Και η οδηγία για τις εκπομπέ, το σύστημα εκπομπών και η οδηγία για τι ανανεώσιμε είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσουμε τον συντονισμό και να μας επιτρέψει, για να επιτρέψει να προχωρήσουμε με το ίδιο βήμα όλοι. Ε, και να υπάρξει ενοποίηση αγορά. Για την ερώτηση του Προέδρου. Φυσικό αέριο ή ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν ξεχνάτε ότι συχνά δίνουμε σημασία, μεγάλη σημασία στο ηλεκτρικό ρεύμα και μικρή σημασία στο φυσικό αέριο. Ε, γιατί κι όμως ε, το αέριο είναι πιο σημαντικό για την ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας. Τώρα, ε, αν κάνουμε τη σύγκριση, οι τιμές που πληρώνουμε εδώ για το φυσικό αέριο είναι πολύ ψηλότερες ε, εδώ από τις ΗΠΑ από ότι η διαφορά που έχουμε στην ε, ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά δεν, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ε, δομή της αγοράς του φυσικού αερίου. Θα πρέπει να δείτε τον ανταγωνισμό, τον αριθμό των φορέων, ε, αν πληρώνουμε δίκαιες τιμές όλοι στην αγορά για το φυσικό αέριο, Τέλο πάντων, όλα αυτά είναι δεδομένα. Είναι πολύ δύσκολο για την Ευρώπη να βρει πόρου ε, κοιτάσματα φυσικού αερίου μέσω, βραχυ, μέσω βραχυπρόθεσμα. Ενώ για το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι το ίδιο. Έχουμε τον ήλιο, το νερό, τον αέρα και επομένως μειώνεται το κόστος. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά, γιατί εμείς στο φυσικό αέριο Πάντα εξαρτώμαστε από το εξωτερικό. Πάντα θα είμαστε πιο εξαρτώμενοι για το φυσικό αέριο από τι αγωγέ από το εξωτερικό. Και αυτέ επηρεάζουν τι εσωτερικέ μα τιμέ. Αλλά μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε στο ηλεκτρικό ρεύμα, ε, κάνοντα τη στροφή προ τι ΑΠΕ, προ ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Ελπίζω αυτό το μήνυμα που ήταν και το βασικό μου μήνυμα να πέρασε. Σας ευχαριστώ και του δύο για του θαυμάσιους λόγου, για τις ωραιότατε απαντήσει στο πρώτο τμήμα τη συζήτηση. το, την πυρηνική ενέργεια ω ενεργειακή πηγή δεν την αναφέρατε καθόλου. Κανένα δεν είπε δύο λόγια. Ε, κάποιος από το, τους ομιλητές, ο κ. Τούρμες, λέει ότι είναι πολύ ακριβή. Δεν ξέρω, δεν λέει ο πρόεδρος. Ε, πάμε τώρα στο δεύτερο πάνελ. Να έρθουν οι ομιλητές παρακαλώ. Ο κ. Τεγκέστ, ο κύριος Σαμαντέρ και ο δόκτωρ Τίλμαν you are coming. Yeah. Well, let me let me invite you to be present with us. We will change our. And now we. Ας έρθουν εδώ στο βήμα παρακαλώ. Ας κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα όμως και να σας ενημερώσω πριν το κάνουμε ότι. To inform about anything, please take a seat. Γίνονται πολλέ φασαρίε, πολλά πηγαδάκια στην αίθουσα. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, Αρχίζουμε με το δεύτερο πάνελ της ακρόασης. Πιλάρ μου, πιλάρ μου, σε παρακαλώ. Πιλάρ μου. Νίκα, Κύριε Νίκα, σας παρακαλώ καθίστε, μην εξαφανιστείτε. Okay, okay. Ε, dear friends, let us start. Please. Τα πηγαδάκια να τα κλείνουμε σιγά σιγά. Θέλω να καλωσορίσω τους ομιλητές του δεύτερου πάνελ Γενικό Διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση ενέργεια ο Ντομινίκ Ριστόρη. Ευχαριστώ που ήρθατε. Στο τέλο τη συνάντηση θα κάνετε μια μικρή ομιλία. Και μην ξεχνάμε βέβαια ότι πάντα όλα όσα λέμε είναι υπό τον έλεγχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό αισθανόμαστε αυτή την ασφάλεια. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ντεγκέστον, ο πρώτο ομιλητής. που είναι από την BASF της Ανβέρσας, από μια εταιρεία χημικών του Βελγίου που την ξέρετε πολύ καλά, που είναι και πρόεδρος της ε, Βελγικής Ομοσπονδίας ε, Χημικών και αντιπρόεδρος μιας ε, οργάνωσης φλαμανδών εργοδοτών και μέλος της Εκλεκτικής Επιτροπής της ε, οργάνωσης των Βέλγων εργοδοτών. Ε, προφανώς είσαστε αρμόδιος να μιλήσετε στο δεύτερο πάνελ για τους χρήστες ενέργειας. Έχετε το λόγο. Είναι πραγματικά προνόμιο το ότι έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι μια εικόνα ενός μεγάλου χημικού εργοστασίου. Το δεύτερο μεγαλύτερο της BASF παγκοσμίω και βρίσκεται στο Βέλγιο, δηλαδή στην Ευρώπη, στη Φλάνδρα όταν σκέφτομαι αυτό το εργοστάσιο και εσεί όταν σκέφτεστε ε, πρέπει να έχετε κατά νου πως πρόκειται για εργοστάσιο που παράγει πάρα πολλά προϊόντα σε ολοκληρωμένε αλυσίδε, αξίες και σημαντικό είναι δύο πράγματα όταν μιλάμε για ενέργεια είναι η αξιοπιστία και η ανταγωνιστικότητα όσον αφορά το κόστος θα επανέλθω στον όρο αυτόν αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να αντιληφθείτε ότι η χημική βιομηχανία είναι μια βιομηχανία όπου η αλυσίδα της αξίας ξεκινάει από τα βασικά προϊόντα, τα πετροχημικά μέχρι τον υψηλότερο βαθμό διήλυσης ε, και επεξεργασίας που βρίσκεται στα φαρμακευτικά προϊόντα. Οπότε ξεκινάμε από το ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια και Άρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η ανταγωνιστικότητα του κόστους. Μια στιγμούλα. Αυτά είναι τα δεδομένα της Eurostat εδώ πέρα. Και βλέπουμε ποια είναι η ζήτηση της βιομηχανίας. Δεν μ' αρέσει να μιλάω για κατανάλωση, να μιλήσουμε για ζήτηση ενέργειας. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα σε αυτό το διάγραμμα πως ολόκληρη η χημική βιομηχανία είναι 11% αλλά 11% παράλληλα αυτά ολόκληρη της ευρωπαϊκής ζήτησης ενέργειας. Αλλά αυτό το οποίο είναι ακόμη σημαντικότερο είναι ότι αυτό το 11% μετά ε, διασπάται ακόμη περισσότερο. Μόλις ένα τρίτο αυτού του 11% έχει σχέση με αυτό το οποίο γενικά λέμε κατανάλωση ενέργειας. Γιατί η χημική βιομηχανία τι κάνει. Τα δύο τρίτα είναι ζωοτροφές, είναι πρώτες ύλες, είναι πρώτες ύλες για δημιουργία αξίας σε τομείς που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και θεωρούνται και σημαντικοί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές αποφάσεις και πράγματι έχουν γίνει οι μελέτες και η Γενική Διεύθυνση ζήτησε μία μελέτη για το που θα είμαστε το 2050, δηλαδή ποια θα είναι η μελλοντική ζήτηση ενέργειας, που θα είναι η ζήτηση ενέργειας και που μπορούμε να εξοικονομήσουμε σε 8 κλάδους έντασης ενέργειας και 4 κλάδους που μπορούμε να ονομάσουμε την ε, τριτογενή παραγωγή. Και βλέπετε εδώ πέρα, και κάτω το οποίο συμφωνεί και με τα δικά μας ευρήματα, ότι η ζήτηση, η ζήτηση ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται στη χημική βιομηχανία. Και γιατί, κυρίες και κύριοι, γιατί η βιομηχανία αυτή κατά 95% δημιουργεί τα απαραίτητα υλικά για όλες τις άλλες βιομηχανίες για την αυτοκινητοβιομηχανία, για την μελλοντική αυτοκινητοβιομηχανία, για μικροεπεξεργαστές. Είτε θέμε να μιλήσουμε για την αιωλική ενέργεια. Οτιδήποτε χρειαζόμαστε τα χημικά συστατικά. Οπότε είναι λογικό ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται η ζήτηση γιατί αυτό βασίζεται στις προβολές της ανάπτυξης. Και νομίζω πως η ανάπτυξη είναι νομίζω αυτό το οποίο θέλουμε στην Ευρώπη. Τώρα, μπορούμε να μιλήσουμε για την ζήτηση της ενέργειας. Σημαντικό για εμάς ως επιχείρηση είναι να πούμε πως ναι, είμαστε επιχείρηση έντασης ενέργειας, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε αυτή την ένταση ενέργειας ή για να αυξήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Εδώ πέρα βλέπετε πώς ο όμιλός μας ε, αντιμετωπίζει το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας παγκοσμίω. Έχουμε παγκοσμίω 27 μονάδες ε, συμπαραγωγής ενέργειας και θέρμανσης. Δηλαδή δεν παράγουμε μόνο ηλεκτρισμό αλλά και θέρμανση γιατί οι χημικές διαδικασίες ε, συχνά μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα θερμότητα την οποία εκμεταλλευόμαστε για να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή αποδετικότητα και να έχουμε τον συνδυασμό ατμού, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν πως 70% του ηλεκτρισμού που χρειαζόμαστε παράγεται σε αυτά τα εργοστάσια τα οποία είναι πάρα πολύ αποδοτικά. Η πρώτη ύλη για αυτά τα εργοστάσια είναι αέριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως η τιμή του αερίου, το ανέφεραν και οι προηγούμενοι ομιλητές, είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς και ένα βασικό στοιχείο του κλάδου μας. Και για την BASF βεβαίως. Παράδειγμα, ένα εργοστάσιό μας στο Λούτβισχάφεν, το μεγαλύτερο εργοστάσιό μας. Για να το αντιληφθείτε, γιατί είναι ίσως κάπως λίγο δύσκολο το διάγραμμα, δύο πράγματα. Έχουμε για εμάς το φυσικό αέριο, το οποίο είναι, όπως είπα, πρώτη ύλη για να φτιάξουμε εκείνα τα μόρια, τα οποία είναι πρόδρομες ουσίες για πάρα πολλά προϊόντα χωρίς τα οποία δεν μπορούμε να ζήσουμε και συνεισφέρουν όπως σας είπα για την παραγωγή και για ολόκληρη την κοινωνία και για το κλίμα μεταξύ άλλων. Παραγωγή παραδείγματος χάρη ε, αμμονίας ε, για 80% του κόστους της παραγωγής ε, αμμονιούχων είναι το φυσικό αέριο. και κάνουμε παράδειγμα τους χάρη μια συμφωνία που μας δίνει 5 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυτό σημαίνει πως έχουμε πολλά εκατομμύρια ως κόστος σε σχέση παραπάνω με τους ανταγωνιστές μας το έτος. Συγκρατήστε αυτό το ένα. Το δεύτερον, στον συνδυασμένο κύκλο, στα εργοστάσια αυτά συνδυασμένου κύκλου που ανέφερα, που κάνουν και τηλεθέρμανση, χρειαζόμαστε και φυσικό αέριο και μετά τι προκύπτει, προκύπτει ατμός από την διαδικασία, αλλά σημασία έχει και το πρώτο μπλε βέλος όπου βλέπετε πως το μεγαλύτερο κομμάτι των αναγκών μας σε θέρμανση προέρχεται από την, πλή, προέρχεται από την πλήρη ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των διαδικασιών. Και έχουμε άρα αυτό το οποίο λέμε Verbund Highly Integrated στα αγγλικά, είμαστε πλήρως ολοκληρωμένοι ως εργοστάσιο. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία ονειρευόμαστε στην Ευρώπη να φτάσουμε ε, γενικώ όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας. Μόνο λοιπόν με αυτό το σύστημα έχουμε εξοικονομήσει 3,4 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα τον χρόνο. Κάτι το οποίο σημαίνει πάνω από ένα εκατομμύριο τόνους ορυκτά καύσιμα το χρόνο. Πάρα πολλά πράγματα λοιπόν κάνουμε όσον αφορά τον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν οι επιχειρήσεις, αλλά όπως και στην μελέτη που παρήγγειλε η Γενική Διεύθυνση, ε, διαπιστώνουμε πως υπάρχουν κάποια όρια σε αυτή τη ε, διαδικασία, οπότε πρέπει να αγοράζουμε ενέργεια από την αγορά. Και περνάμε άρα στο επόμενο και αυτό είναι σημαντικό να δείτε αυτή την εικόνα. Ναι. Βάλτε το σπάρκαλο σε πλήρη οθόνη. Τι βλέπουμε λοιπόν. Ότι μιλάμε πολύ για τις τιμές της αγοράς. Αλλά υπάρχει διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και κόστους. Και αυτό το οποίο μετράει για μας είναι το συνολικό κόστος. Δεν είναι η τιμή της αγοράς. Γιατί πράγματι δεν νομίζω πως μπορεί κανείς να φέρει αντίρρηση πως η τιμή της αγοράς μέσω των προσπαθειών της Ευρώπης και των πρώτων βημάτων απελευθέρωσης της ε, αγοράς πράγματι έπεσε. Δεν έχουμε φτάσει βεβαίως στην εναρμόνιση, αλλά διαπιστώνουμε πως οπωσδήποτε υπάρχει μια κάποια αποσύνδεση και μια μείωση. Στο Μπενελούξ, Γαλλία, Γερμανία, γιατί, γιατί ακόμα δεν είναι τέλεια η αγορά του πετρελαίου. Δηλαδή το όνειρο της Ευρώπης για μια ενεργειακή αγορά όπου τα πάντα ρέουν χωρίς ε, φραγμούς ε, είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει αλλά ε, δεν, αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχουν διασυνδέσεις και τέτοια πράγματα. Αλλά το ότι πέφτουν οι τιμές αγοράς είναι η μία πτυχή, αλλά κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το κόστος. Ανεβαίνουν τα κόστη του δικτύου, φόροι και τέλη ανεβαίνουν και ανεβαίνουν τόσο πολύ ώστε αντισταθμίζουν και με το παραπάνω το ότι πέφτουν οι τιμές της αγοράς. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι ίσως η τιμή της αγοράς πέφτει, αλλά αυτό είναι αδιάφορο για μια επιχείρηση. Για μια επιχείρηση μετράει μόνο το τι πληρώνει. Και επανερχόμαστε εδώ πέρα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να κρατήσουμε το κόστος υπό έλεγχο. Βεβαίως θα συνεχίσουμε τους ε, στόχους μας. Έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους. Ε, ως BSF 2020 θέλουμε να έχουμε μία μείωση κατά 40%. Όταν μιλάμε λοιπόν για το κόστος ε, της ενέργειας, μην ξεχνάμε πως έχουμε 1,8 δισεκατομμύρια που ρίχνουμε στην έρευνα και το 1 τρίτο από αυτά πηγαίνουν την έρευνα για την ενέργεια. Χωρίς αυτό δεν θα έχουμε καλύτερα αυτοκίνητα, χωρί δεν θα έχουμε καλύτερες μπαταρίες, αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας κτλ. Όλα αυτά λοιπόν σχετίζονται με την καινοτομία και βεβαίω μετά με την φορολογία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Πολύ πλήρη η ομιλία σας, πολύ ξεκάθαρη οι απόψη σας. Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος, τις τιμές ενέργειας, και τα ενεργειακά γενικώ θέματα. Να δώσω τώρα το λόγο στον δεύτερο μιλητή, τον κύριο Σαντζέι Ζαμαντάρ. Από την Πεντζάμπ. Και στο ΕΛΕΣΥ e και χημική μηχανολόγια και χημικός μηχανικός ήταν στην Αρσελόρ Μιτάλ, αρχικά στην Ουρμανία και τώρα είναι αντιπρόεδρος στην Ευρώπη. Στην Αρσελόρ Μιτάλ πάντα. And Arcelor Mittal Ostrava. So we Άρα από τη χημική βιομηχανία πήγατε στη Χαλιβουργία. Κύριε Σαμαντάρ, Thank you, uh, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Director General. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές. Πραγματικά είναι προνόμιο για μένα να σας παρουσιάσω τις απόψεις ε, του κλάδου της Χαλιβουργίας ό,τι αφορά την ενέργεια και το ETS. Και πολλά από όσα πω σήμερα εδώ ε, θα είναι εκ μέρους ε, των παραγωγών χάλιβα από την Ανατολική κυρίως Ευρώπη. Να σας δώσω αρχικά κάποια βασικά στατιστικά στοιχεία να δούμε τη σημασία της χαλιβουργίας για την οικονομία στην Ευρώπη. Προφανής η σημασία ε, είναι δύσκολο ίσως να διακρίνεται τη διαφάνεια ε, σε όλα τα στοιχεία, αλλά βλέπετε ότι κυρίως ε, οι θέσεις εργασίας είναι το βασικό, 330.000 περίπου. Φυσικά έχουμε ε, μείωση 25% και στις εκπομπές ε, διοξιδίου από το 1990 και είναι και ένας στόχος που εξακολουθεί να είναι πρωταρχικός για να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές ε, του κλίματος. Ποιες είναι οι βασικές ανησυχίες στον κλάδο. Το 20% μείωση στην απασχόληση από το 7 και μετά, η μείωση 28% της ζήτησης χάλιβα το 14 σε σχέση με την αφετηρία το 7 και από την ανακαμψή ωφελούνται οι ε, εισαγωγές. Από την άλλη πλευρά έχουμε υψηλές τιμές ενέργειας και αθέμητες εμπορικές πρακτικές από χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη είναι η οικονομική μόχλευση του τομέα της χαλιβουργίας για την κοινωνία. Βλέπετε γιατί πρέπει να παραμείνει βιώσιμος αυτός ο κλάδος. Από στατιστικής πλευράς στα, στατιστικής πλευράς, Εάν έχουμε πρόσθετη ζήτηση της τάξης ενός ευρώ για προϊόντα χάλιβα, έχουμε 3,1 ευρώ, τα 2,1 πηγαίνουν στους άλλους προμηθευτές. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται και ε, η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠΑ. Ένα πρώτο στοιχείο ε, υποστήριξης που χρειαζόμαστε. Το ενεργειακό κόστος. Βλέπετε μια πολύ ανησυχητική τάση σε ό,τι αφορά το μερίδιο στην αγορά εξαγωγών για ενεργοβόρα αγαθά. Βλέπετε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη μείωση. Και αυτό μας ανησυχεί. Και αυτή την τάση θα πρέπει να αναστρέψουμε. Γιατί θέλουμε να πετύχουμε την επανεκβιομηχάνηση της Ευρώπης. Αυτός είναι ο στόχος. Βλέπετε τώρα δύο γραφήματα. Σε αυτά βλέπετε ότι το ενεργειακό κόστος ήδη είναι ένα τεράστιο κομμάτι από το περιθώριο, ε, από τα περιθώρια των εταιριών χαλιβουργίας. Έχουμε την ανάγκη να καταστήσουμε όλους αυτούς τους ενεργοβόρους τομείς, μεταξύ αυτών και τη χαλιβουργία, ενεργειακά πιο αποδοτικούς. Έχουμε να, ε, να λύσουμε τα εξής τρία προβλήματα. Πώς θα έχουμε ισότιμο παιδί ανταγωνισμού με άλλου ανταγωνιστέ όταν αυξάνονται οι ενεργειακοί φόροι και οι Δεύτερον, θέλουμε μεγαλύτερη ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς, δηλαδή να προωθήσουμε την ανταπόκριση στη ζήτηση και υπάρχουν και αυτοί οι μηχανισμοί δυναμικότητας που πρέπει να εξετάσουμε και έχουμε και το σύστημα ETS ε, που είναι αμφισβητήσιμο και πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τα κίνητρα για την απαλλαγή από τον άνθρακα. Έρχομαι τώρα σε κάποια άλλα. Είπαμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ανταγωνιστικότητα λόγω πολλών δασμών, φόρων, ιδίως ό,τι αφορά ε, την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ε, υπάρχουν διάφορα προγράμματα, διάφοροι μηχανισμοί και αυτό δημιουργεί ένα μη ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού και δημιουργεί προβλήματα στον κλάδο. Πώ θα καταλήξουμε όμω να έχουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, κυρίω κατά την άποψή μας τουλάχιστον, χρειάζονται δύο δέσμες δράσεων. Πρώτα απ' όλα εξαιρέσεις ε, για να έχουμε τις κατάλληλες τιμές ενέργειας και δεύτερον να έχουμε σύγκληση ε, των φόρων και δασμών σε επίπεδο κρατών μελών. Κάτι που δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή, τη σύγκληση αυτή δηλαδή. Τρίτο σημείο. Θέλουμε να έχουμε την ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας. Αυτοί οι μηχανισμοί δυναμικότητας μπλοκάρουν ε, την ανάπτυξη της αγοράς και κατά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως έσχατη λύση. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει το κίνητρο της δίκαιης αμοιβή. Έρχομαι στο άλλο σημείο που μας ανησυχεί, το ETS, όπως προτείνεται και ισχύει αυτή τη στιγμή επηρεάζει τη χαλιβουργία το Not ΝΑΤΦΟΡ. Για την επίτευξη των στόχων του ETS σχεδιάζει να επιτρέψει πληστηριασμό του 57% των δικαιωμάτων η Κομισιόν, οδηγώντας στην απαλλαγή από το άνθρακα για κάποιε χώρε. Και θέλει με αυτό να πετύχει και κάποια έσοδα. Δημιουργεί όμως κάποια τεχνητά benchmarks και αυτό στρεβλώνει την κατάσταση για πολλούς ενεργοβόρους τομείς. Και ποια είναι η συνέπεια. Και η αλυσίδα αξίας ε, σε πολλά κομμάτια της ε, και πολλές τέσσερα. Σας θα χαθούν. Κατάγομαι από την Ανατολική Ευρώπη και πρέπει να σας πω ότι εκεί ε, θα πλήξει πιο πολύ και καταρχάς αυτή η προσέγγιση, αυτό το μέτρο. Ποια είναι τώρα η προβλεπόμενη επίπτωση ο αντίκτυπος ε, του ETS ε, μετά το 2020 στη Γαλλιμπουργία. Έχουμε μία μελέτη που τη βλέπετε, δείχνει ότι τέσσερις θα είναι οι βασικές αρνητικές συνέπειες. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε έλλειψη 48% σε ό,τι αφορά το free allocation. Το 2030 76% του άμεσου κόστους δεν θα αντισταθμιστεί, με αποτέλεσμα να έχουμε 34 δις ευρώ παραπάνω κόστος για την περίοδο στο 2030. 28 ευρώ, α, ανά ε, τόνο χάλιβα. Πολύ ανησυχητικά στοιχεία. Τώρα κύριε Πρόεδρε, γιατί εμείς λέμε ότι το σχέδιο ETS ε, στη σημερινή του μορφή είναι αντιπαραγωγικό σε ό,τι αφορά κίνητρα για το κλίμα. Τα ορυκτά καύσιμα δεν θα ορίζουν πλέον τις τιμές, κατά την άποψή μας, Ούτε είναι ωραίο να έχουμε μια προσέγγιση, ένα μέγεθος για όλους. Είναι λίγο επικίνδυνο, μάλιστα. Γιατί θα δώσει τη δυνατότητα ίσως ε, σε διαρροές άνθρακα ή σε κάποια άλλα ε, Και θα υπάρξουν και ελλείψεις. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Δεν υπάρχει λοιπόν κίνητρο να επενδύει κανείς σε καινοτόμες τεχνολογίες για να στηρίξει τους μηχανισμού αλλαγής κλίματος. Εμείς όμως θέλουμε παρόλα αυτά να επενδύσουμε σε αυτό. Έτσι, οι διαπραγματεύσει ε, για το ETS ενδέχεται να μην λύσουν τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τι απαιτείται λοιπόν, αυτό το 57% ε, όγκο των πληστηριασμών πρέπει να μειωθεί κατά 5,5% αλλά να ξεκινήσει από ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο, θα έλεγα 49%. Θα πρέπει να αλλάξουν εντελώς ε, τα benchmark και αυτό να βασίζεται στις μονάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή χωρίς τεχνητές επίσχες μειώσεις ή πλεονάσματα. Και ε, το μη κινδύνου όπως ε, ο Χάλιβας θα πρέπει να παίρνουν ε, free allocation της τάξης στο 100% θα πρέπει να έχουμε πλήρη αντιστάθμιση για το διοξίδιο και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνουν με τις μη τα μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα. Αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιείται για ελεύθερη διάθεση. Παρόλα αυτά, πολλά, ε, πολλές μονάδες μπορεί να χρειαστεί να κλείσουν λόγω του πολύ σημαντικού ε, έξτρα κόστους. Τώρα, για το σχέδιο του ETS μετά το 2020 θα εξαγάγει, πιστεύουμε, θέσεις εργασίας και θα εξαγάγει άνθρακα. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία αξίζει να μπορούμε να επενδύσουμε στις μονάδες, να γίνουμε ε, πρωταγωνιστές σε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε υποστήριξη. Πρώτα απ' όλα, ένα ανταγωνιστικό σωρευτικό ενεργειακό κόστος, είναι ένα κριτήριο, είναι μια προϋπόθεση και δεύτερον να έχουμε ένα διάλογο για το ETS για να μην έχουμε ε, διαρροή άνθρακα μετά το 2020. Μπορεί για κάποιους να μην θεωρείται ε, ζήτημα ανησυχίας προς το παρόν. Εμείς όμως μιλάμε για μετά το 2020. Θέλουμε λοιπόν ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού ε, για το χάλιβα στην Ευρώπη. Για να πετύχουμε πέντε βασικούς μας στόχους, να διατηρήσουμε την απασχόληση. Σας είπα πριν ότι έχουμε 330.000 θέσεις εργασίας, αλλά σας είπα ότι μειώθηκαν θέσεις αυτές από το 7 στο 14. Σας είπα επίσης για το 1 ευρώ που οδηγεί σε 3,1 σε άλλες ε, εφοδιαστικές αλυσίδες. Τρίτον, θέλουμε περισσότερη ενεργειακή ε, ασφάλεια, θέλουμε να επενδύσουμε ε, στη γενοτομία και πέμπτον, εξίσου σημαντικό, να βελτιώσουμε την αλλαγή του κλίματος για το κοινό μας όρεμα για την Ευρώπη. Από κοινού πιστεύω μπορούμε να βρούμε ανταγωνιστικές λύσεις, γιατί το βασικό είναι να μην χάσουμε σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας και μειωθεί η ανταγωνιστικότητά μας. Είπε ο Επίτροπος ότι υπάρχουν κάποιες δράσεις ε, που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα. Η δική μας συμβολή και για το ETS είναι αυτή που μας σας παρουσίασε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα τα νούμερα που μας δώσατε για τους διάφορους κλάδους. φτάσετε σε ανάλογα συμπεράσματα με προλαλήσαντες. Και τώρα πάμε στη χημιακή βιομηχανία. Ο τρίτος ομιλητής είναι ο κύριος Τίλμαν, ο δόκτωρ Τίλμαν. Από το Βερολίνο. Βιολόγος στο Πανεπιστήμιο Φραγκφούρτης και Κίλ. Αυτά έχετε σπουδάσει. έχετε μια πολύ ψηλή θέση σε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο στη Γερμανία. Και δουλεύετε κι εσείς για την ΠΑΣ ως διευθυντής του Συμβουλίου των Χημικών Βιομηχανιών. Και τώρα είσαστε Διευθυντή Οργάνωση Γερμανικών Χημικών Βιομηχανιών. Θέλουμε να σας ακούσουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στη μεγάλη βελική βιομηχανία, την BASF και στη γερμανική βιομηχανία που γνωρίζετε τώρα. Να δούμε αν υπάρχουν διαφορές στο κόστος της ενέργειας στο Βελίο και στη Γερμανία. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Γενική Διευθύντα. Τώρα δεν θα κάνω εγώ συγκρίσεις μεταξύ των διαφορετικών ε, βιομηχανιών. Θα μιλήσω για τη χημική βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα και το κόστος ενέργειας. Η χημική βιομηχανία είναι ο κλάδος εκείνος με το υψηλότερο κόστος της ενέργειας και την υψηλότερη ζήτηση ενέργειας. Ήδη αναφέρθηκε η σημασία που έχει για εμάς γιατί Βεβαίως ε, είναι πρώτη ύλη, αλλά τη χρειαζόμαστε και για την παραγωγή. Οπότε είναι διπλό το θέμα της ανταγωνιστικότητας των τιμών της ενέργειας για εμάς. Αυτά πρέπει να τα έχουμε πάντα κατά νου, είναι πολύ σημαντικά. Αν δείτε λοιπόν το κόστος και τις ποσότητες εδώ πέρα τους όγκους, βλέπετε πως μονάχα στο ρεύμα στη Γερμανία έχουμε μια κατανάλωση η οποία ανταποκρίνεται σε 10 εκατομμύρια τετραμελή ε, νοικοκυριά. Ένα ε, τεράστιο δηλαδή ποσοστό του ε, πληθυσμού, μισός πληθυσμός θα έλεγα. Οπότε με τα προϊόντα αυτά θα έλεγα πως εμείς στην πλάτη μας κουβαλάμε το βάρος ενέργειας και διοξιδίου του άνθρακα για όλους ή τέλος για πολλούς Κλάδου τη βιομηχανία, γιατί εμεί βάζουμε την ενέργεια στα προϊόντα τα οποία οι άλλοι τα αγοράζουν έτοιμα και παράγουν προϊόντα υψηλή απόδοση για να φτιάξουν παραδείγματο χάρη φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, αυτοκίνητα, υπολογιστέ, κτίρια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε αν δεν βάζαμε εμεί αυτή την ενέργεια μέσα στα προϊόντα δεν θα μπορούσαν όλοι οι υπόλοιποι παρακάτω στην αλυσίδα να φτιάξουν προϊόντα υψηλή απόδοση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είναι σημαντικό για εμάς να βλέπουμε την συνολική εικόνα σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και δημιουργίας αξίας και όχι μόνο να βλέπετε τη χημική βιομηχανία μεμονωμένη. Αν δούμε τώρα την χημική βιομηχανία βλέπουμε πως είμαστε βεβαίω ε, πάρα πολύ ενεργοβόρος βιομηχανία. Βλέπετε όμως ότι χρησιμοποιούμε λιγότερη ενέργεια. Βλέπετε πόσο αποδοτικά χρησιμοποιούμε την ενέργεια. Η πάνω γραμμή δείχνει την εξέλιξη της παραγωγής μας από το 1990 η οποία αυξήθηκε κατά 60% και η κάτω-κάτω γραμμή μας δείχνει πώς έχει μειωθεί η ειδική κατανάλωση ενέργειας. Οπότε η ενεργειακή μας αποδοτικότητα μεταξύ 1990 και σήμερα έχει διπλασιαστεί πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα. Οπότε με όλες τις προσπάθειες που κάνουμε νομίζω πως αξίζει η ενεργειακή αποδοτικότητα γιατί χρησιμοποίησαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Θα μπορούσε βέβαιως να ρωτηθεί κανείς ποια είναι η κινητήριος δύναμη για την ανταγωνιστικότητα σε σχέση με την ενέργεια. Είναι βεβαίως η τιμή του ρεύματος είναι οι τιμές των πρώτων υλών και όλες οι πρώτες που χρησιμοποιούμε, που απο... τα βασικά χημικά στοιχεία τα οποία έχουν τιμές παγκόσμιας αγοράς. Δηλαδή βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο ανταγωνισμό με τα προϊόντα μας και πρέπει παρόλα αυτά να πληρώσουμε ψηλότερες τιμές ενέργειας και πρώτων υλών για να φτιάξουμε αυτά τα προϊόντα. Αυτή είναι η βασική διαφορά λοιπόν και βεβαίως στην Ευρώπη έχουμε λίγους φυσικούς πόρους και έχουμε πολύ ρυθμισμένη αγορά. Οι δύο καμπύλες αυτές μπορώ να σας εξηγήσω πάρα πολύ εύκολα. Η μία πλευρά είναι αέριος, την άλλη πλευρά είναι οι τιμές του ρεύματος Έχουμε λοιπόν βλέπετε σαφή διαφορά όσον αφορά τις τιμές ε, του αερίου. Αναφέρθηκε ήδη τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε την τιμή του αερίου. Ένα πάρα πολύ απλό μπορούμε να κάνουμε fracking ε, υδρορογμάτωση στην Ευρώπη και έτσι θα έχουμε αυτομάτως πολύ μεγαλύτερη παραγωγή αερίου και θα μειωθεί η τιμή του. Τουλάχιστον ε, διπλάσια ή τριπλάσια, γιατί είναι η τιμή αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις ΣΥΠΑ. Στο ρεύμα βλέπετε ξεκάθαρα έχει αυξηθεί η τιμή για την βιομηχανία. Ψέματα, ψέματα λέει ο κύριος Τούρμες. Πα, τι είναι αυτά που μας δείχνετε τα στατιστικά στοιχεία. Α, μα έχετε κι άλλα ευχαριστώ, λέει ο, ο μιλητής για την τιμή του ρεύματος πρέπει να κάνουμε σαφή διάκριση. Είναι τιμή του ρεύματος που κοιτάμε μόνο την ε, τιμή, όπως είπαμε, της αγοράς και αφαιρούμε όλα τα άλλα. Μα στη χημεία σας είπα αυτό δεν απαλλάσσονται ούτε 10% των επιχειρήσεων. Όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουν την πλήρη τιμή. Μην μου λέτε λοιπόν ότι είναι ψέμα, είναι η αλήθεια και αν συγκρίνετε τις τιμές του ρεύματος θα δείτε πως σε σχέση με τη ΣΥΠΑ πληρώνουμε την διπλάσια τιμή στη Γερμανία. Και για να το ξεκαθαρίσω, ε, έχουμε εδώ πέρα μια δημοσκόπηση μεταξύ των ε, μελετών μας, όπου κάνουμε μια σύγκριση των διαφόρων ε, σημείων παραγωγής. Και βλέπετε πάνω-πάνω την Γερμανία Και μάλιστα δεν μιλάμε για τιμή αγοράς. Βλέπετε το τι πληρώνουν οι γερμανικές εταιρείες στη Γερμανία και το τι πληρώνουν σε άλλες σημαντικές ανταγωνιστικές περιοχές του κόσμου. Βλέπετε παραδείγματο χάρη στη ΣΥΠΑ ή στην Κίνα. Ας δούμε μόνο αυτές τις δύο. Και πάλι βλέπετε ότι είμαστε σε διπλάσιο επίπεδο, γιατί αυτοί αν θέλετε έχουν τη μισή τιμή από αυτό το οποίο πληρώνουμε στη Γερμανία. Οπότε, στην Γερμανία έχουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα, μειονέκτημα και είναι αδιάφορο το εάν ε, συμπεριλάβω την απαλλαγή που μου λέτε εσείς ή όχι. Το ερώτημα λοιπόν. Το ζήτημα το οποίο συζητήθηκε στο πάνελ για το εάν μπορούμε να συνδυάσουμε την παραγωγή με την παραγωγή ρεύματος. Μα αυτό είναι τελείως αντιαποδοτικό. Οι, τα εργοστάσια μας λειτουργούν συνεχώς. Αν τα αναβοσβήνουμε, θα είναι πολύ περισσότερες οι εκπομπές. Είναι καλές αυτές οι ιδέες αλλά δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα. Ουδεμία. Οπότε δεν είναι, είναι απαράδεκτα αυτά. Το επόμενο. Να δείτε το ρυθμιστικό βάρος, πώς ε, αθρίζεται το κόστος. Το είπαν και οι συνάδελφοι, βλέπετε τη σύγκριση είπα, Γερμανίας. Έχουμε μια ελαφρώς καλύτερη θέση όσον αφορά την ε, παραγωγή του κόστους ε, και το δίκτυο. Έχουμε σαφώς ε, υψηλότερα τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και βεβαίως πανευρωπαϊκά έχουμε την επιβρόστιη επιβάρυνση του εμπορίου εκπομπών. Όλα αυτά σας δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η διαφορά της ανταγωνιστικότητας για τη χημική βιομηχανία παραδείγματο χάρη μεταξύ Γερμανίας και ΕΙΠΑ. Και το κενό που βλέπετε, το χάσμα αυτό, είναι αυτό το οποίο πρέπει να καλύψουμε. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό μας μειονέκτημα και πρέπει να το καλύψουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Αυτό αντιμετωπίζουμε στην κοινική βιομηχανία. Λοιπόν, έχω τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα πως οι επενδύσεις στη Γερμανία βλέπετε είναι η μπλε γραμμή, ε, δεν κινούνται σχεδόν καθόλου. Η άλλη γραμμή είναι οι επενδύσεις γερμανικών εταιριών στο εξωτερικό. Τι μας δείχνει αυτό, πως έχουμε σαφείς ε, αυξήσεις ε, των επενδύσεων στο εξωτερικό, ειδικά με το σχιστολιθικό αέριο. Ποιο είναι το κίνητρο. Βεβαίως η αγορά αλλά εάν δείτε το, την πάνω πάνω στήλη βλέπετε πως στις ΙΠΑ οι περισσότερες επενδύσεις μιλάμε πάντα για ενεργοβόρες βιομηχανίες πηγαίνουν εκεί γιατί είναι τόσο φτηνή η τιμή της ενέργειας. Οπότε αν δούμε το που βρίσκεται η ανταγωνιστικότητά μας σήμερα μπορώ να πω πως έχουμε το υψηλό κόστος που δεν αλλάζει, έχουμε δεύτερον ένα σαφές μειονέκτημα στην ανταγωνιστικότητα απέναντι σε περιοχές όπως είπα. Τρίτον, έχουμε μια σαφώς χειρότερη θέση όσον αφορά το κόστος σε σχέση με το εμπόριο εκπομπών και όλες αυτές τις πολιτικές για το κλίμα και σήμερα βλέπουμε διαρροή επενδύσεων προς τη ΣΥΠΑ ήδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. σαφέστατο και ηχηρό το μήνυμα, ακόμα πιο ηχηρό σε σχέση με το προηγούμενο από το Βέλγο εκπρόσωπο. Δύσκολο ήταν το πλαίσιο με στο οποίο κάνατε την παρέμβασή σας και τώρα πάμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο κύριος Πίπερ από το ΕΛΚ. Ja, ich möchte zunächst eine... Θα να σχολιάσω ένα διάγραμμα εδώ πέρα που εξαιρέτησε τον κύριο Τούρμες ε, όπου ήθελε να μας πει στο τέλος του πρώτου πάνελ ότι θα αν καταργούσαμε τις ειδικέ ε, τιμές για τους βιομηχανικούς πελάτες οι μεσές επιχειρήσεις θα είχαν χαμηλότερες τιμές. Ήταν λοιπόν ένα διάγραμμα το οποίο χειραγωγούσε τα πράγματα γιατί ακόμα και αν καταργούσαμε τις ειδικές τιμές ε, θα είχαμε μόνο ένα κλάσμα της ε, χαμένης ανταγωνιστικότητας σαν οπότε η βιομηχανία εκδιώκεται από την Ευρώπη. Λοιπόν, έχω ένα ερώτημα και στους τρεις να απευθύνω. Ήταν ε, εντυπωσιακά αυτά τα στατιστικά στοιχεία που μας δείξατε για τις τιμές της ενέργειας ε, και το βάρος που κουβαλάτε εσείς για τις άλλες βιομηχανίες. Θα ήθελα να μάθω πώς έχουν οι επενδύσεις τώρα στον κλάδο του καθενός σας. Πού επενδύεται, σε ποια μέρη του κόσμου, ποιες χώρες είναι οι στόχοι σας και σε ποιο βαθμό έχετε νέα ε, εργοστάσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Νταν Νίκα, Σοσιαλδημοκράτες. Ε, ε, ευχαριστώ. Καταρχάς, θέλω να πω στους προσκεκλημένες μας ότι σε ό,τι αφορά την προστασία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αυτό είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Και δεν θέλουμε καθόλου να εξάγουμε θέσεις απασχόλησης και να εισάγουμε προφανώς εκπομπές διοξείδιο του άνθρακα. Θα ήθελα λοιπόν να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις με βάση την εμπειρία που έχω από τη Ρωμανία, τη χώρα μου. Δεν ξέρω πολλά για τη χημική βιομηχανία γιατί 7 από τα 8 χαλιβουργικά εργοστάσια που υπήρχαν στη Ρουμανία έκλεισαν πέρυσι. Ελπίζω όμως ότι με τη νέα πολιτική της Κομισιόν για το Φυσικό Αέριο θα ξανανοίξουν και οι τιμές θα είναι τιμές αγοράς. Ξέρω όμως το χαλιβουργικό ε, κλάδο. Είμαι από τον Καλάτσι στην Ρουμανία και ένας από τους ομιλητέ μας, μας είπε ότι υπήρχαν κάποτε 40.000 εργαζόμενοι εκεί. Σήμερα υπάρχουν 7.000. Κάτι που δεν καταλαβαίνω καλά. Ποια είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πριν από τρία χρόνια ε, ήμουν στο Υπουργικό Συμβούλιο της Κυβέρνησης και ε, ρώτησα αν μπορούμε να βοηθήσουμε τον κλάδο ε, μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η Κομισιό μου είπε ότι ο κλάδος αυτός δεν χρήζει βοήθειας. Πώς μπορούμε να κρατήσουμε τις ε, θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει τουλάχιστον να βγάζουν τα προστοζήν. Ε, και για, για να βγάζουν τα πεστοζήνη θα πρέπει να έχουν θέσει απασχόληση, αλλά οι βιομηχανίε θα πρέπει να μην έχουν χασούρα. Για το ETS, αυτή τη στιγμή, μετά τη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας εκπομπών, δεν υπάρχει μία χαλιβουργία στην Ευρώπη που μπορεί να σεβαστεί αυτού τους κανόνες. Επίσης, Υπάρχει κανένα, κάποιο εργοστάσιο της, με, της ΕΜΕΤΑΛ, τη ε, χαλιβουργικής αυτής εταιρείας που εκπροσωπείτε. Ε, υπάρχει λοιπόν κάποιο εργοστάσιο που μπορεί να σεβαστεί τους τι ETS. Τρεις ε, σύντομες ερωτήσεις. Θα ήθελα το πάνελ να μου απαντήσει μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Αλλά ποιο είναι το κόστος ενέργειας στο συνολικό κόστος της παραγωγής. Γιατί ε, Διερωτώ είναι 5, 10, 15, 20, 60. Γιατί αν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα, θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το σχετικό βάρος της ενέργειας στο συνολικό κόστος παραγωγής. Δεύτερη ερώτηση για το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Θα γίνει μια μεγάλη συζήτηση και στην Επιτροπή μα και γενικά στο Κοινοβούλιο και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να βρούμε το σωστό συμβασμό ούτε για τον τομέα τη ενέργεια, ούτε για τη βιομηχανία γενικά, ούτε για να μπορέσουμε να αφήσουμε τελικά την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Τι θεωρείτε ότι είναι ε, μια δίκαιη τιμή για το διοξείδιο του άνθρακα και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τις ε, δομές για τη διαρροή του διοξείδιου του άνθρακα στο σύστημα ETS. Για το τελευταίο slide του κ. Μπιχέστ που αναφέρθηκε στην καινοτομία. Ξέρω ότι οι βιομηχανίες σας είναι ε, βιομηχανίες που επενδύουν στην καινοτομία πάντα αλλά επενδύεται στην κυκλική οικονομία. Άκουσα τη λέξη Φερμπούντ, όπου είπατε ότι η ενσωμάτωση των διαφόρων συνιστοσών είναι σημαντική, αλλά πώς επενδύεται στην ε, κυκλική καινοτομία. Υπάρχει καινοτομία εκεί για να αποθηκεύουμε το διοξείο του άνθρακα και να το ξαναβάζουμε δηλαδή στο κλασικό κύκλο παραγωγής της βιομηχανίας σας. Ο κύριος Τούρμες από τους Πράσινους. ενδιαφέρον. Έχουμε ακαδημαϊκούς εδώ, που είναι ουδέτεροι και που δείχνουν Εγώ δεν κάλεσα κανένα από τους δύο μιλητές. Έχουμε δύο ακαδημαϊκούς που δείχνουν ότι σήμερα για το ηλεκτρισμό οι ενεργοβόρες ε, επιχειρήσεις που εσείς εκπροσωπείτε μέσω των ανεώσιμων συν χαμηλών τιμών χοντρικής, συν εξαιρέσεις και μια σειρά από άλλα πράγματα ε, μέσω των αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις κτλ. Έχετε τιμές που είναι πολύ κοντά στις τιμές χοντρικής και τώρα δείχνετε εσείς Γερμανοί μια γραφική παράσταση όπου λέτε ότι η τιμή είναι τριπλάσια ή πενταπλάσια ας πούμε από τι είναι. Ως ε, Εμεί είμαστε μεταξύ των ακαδημαϊκών και των λομπιστών. Και είμαστε νομοθέτες. Τι επιλογή να κάνουμε. Πείστε με. Ότι μας δείξετε τα πραγματικά νούμερα. για να μπορέσουμε πραγματικά να δούμε αν έχετε εσείς δίκιο ή αν έχουν δίκιο οι ακαδημαϊκοί. Τώρα, τρεις ερωτήσεις προς τον εκπρόσωπο της Μετάλ. Στην εταιρεία σας κερδίσατε 400 εκατομμύρια ευρώ από τη δεύτερη και τρίτη φάση του ETS. Η εταιρεία σας επίσης αγοράζει διεθνείς, ε, διεθνή δικαιώματα, αγόρασε μάλλον διεθνή δικαιώματα ETS. Το δεύτερο εξάμεινο του 2012 αγοράσαμε πληρώνοντα 0,5 ευρώ τον τόνο ε, δισεκατομμύρια ε, δικαιώματα εκπομπών. Έτσι κάνετε αντιστάμιση του κινδύνου, όχι μόνο μέχρι το 2020, αλλά και μέχρι το 2020. Έχετε και επιστοποίηση για κάτι τέτοιο. Και μια ακόμα ερώτηση. Η χαλιβουργική εταιρεία Κόπει ο πρόεδρος του ομιλητή. Η κυρία Νίμπλερ. very sorry. Time is over. Τελείωσε ο χρόνος σας κύριε Τούρμες. Κυρία Νίμπλερ. Äh, σας ευχαριστώ. Μου ευχαριστήσω και τους τρεις ομιλητές. Πολύ ενδιαφέροντες. Λοιπόν, Πρώτη ερώτηση. Ο κύριος Τίλμαν αναφέρθηκε στα όσα είπαν οι προλαλήσαντες στο πρώτο πάνελ. Θα ήθελα να ακούσω και από τους τρεις ομιλητές για το πρώτο πάνελ. Τι άποψη έχετε. Και να τα ανακατέψουμε λίγο την επόμενη φορά τα πάνελ, κύριε Πρόεδρε. Να έχουμε μια καλύτερη συζήτηση. Δεύτερη ερώτηση. Ενεργειακή αποδοτικότητα μας είπατε από το 90 μέχρι το 2015 την έχετε διπλασιάσει. Ε, τότε γιατί να σταματήσει αυτή η διαδικασία, γιατί να μην συνεχιστεί. Γνωρίζω πως υπάρχουν κάποια όρια που καθορίζει η φυσική, αλλά που αφού ήσασταν τόσο φιλόδοξοι τα προηγούμενα χρόνια, γιατί να μην συνεχίσετε. Επόμενη ερώτηση, διοξίδιο του άνθρακα, το ανέφερε ο συνάλφος, έχουμε αυτή τη στιγμή χαμηλή τιμή ρήπου. Υπάρχει περιθώριο νομίζω να ανέβει, αλλά το θέμα είναι τι θεωρείτε εσείς ότι είναι οικονομικά ανεκτό και μετά στον εκπρόσωπο της Χαλιβουργίας. Υποθέτω πως η Χαλιβουργία βεβαίως έχει και προβλήματα λόγω της ανάπτυξης της ε, Κίνας, ε, του τεράστιου ανταγωνισμού από την Κίνα. Είχαμε και εδώ πέρα την συζήτηση για το καθεστώς οικονομίας της αγοράς για την Κίνα και τις υποχρεώσεις ε, του ΠΟΕ αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μήπως αυτό είναι σοβαρότερο πρόβλημα για εσάς από ότι το πλαίσιο της εμπορία εκπομπών. Σας ευχαριστώ. Και τώρα οι μιλητές μας μπορούν να απαντήσουν. Με αντίστροφη σειρά. Ξεκινάμε από το την BASF, Γερμανία, μετά Χαλιβουργική Εταιρεία και μετά τελειώνουμε με την BASF του Βελγίου. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, για τις επενδύσεις, κύριε Πίπερ, ήταν αυτό ακριβώς που ήταν το διάγραμμα. Οι επενδύσεις στη Γερμανία είναι απλά συντήρηση των εγκαταστάσεων, δεν χτίζονται νέα μεγάλα εργοστάσια όλες οι μεγάλες εγκαταστάσεις έντασης ενέργειας κατά κανόνα χτίζονται εκτός Ευρώπης, εκεί όπου είναι φτηνή η ενέργεια. Κυρίως είπα, όπου χτίζονται σήμερα τέτοια εργοστάσια, γιατί είναι τόσο φτηνό το ρεύμα και το σχιστολιθικό αέριο. Επίσης, ε, το... Ε, η πολυ το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ φθηνότερο και χρειαζόμαστε, όπως σας είπα, πάρα πολύ ηλεκτρικό ρεύμα για να παραχθεί. Μετά, επόμενο ερώτημα, νομίζω απευθυνόταν προς την ε, Κομισιόν, δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα για την ε, Ρουμανία. Μετά με ρωτήσετε για το συνολικό κόστος των επενδύσεων. Όχι. Με ρωτήσετε για το συνολικό κόστος και την κυκλική οικονομία. Για την χημική βιομηχανία είναι το ψωμοτήρι μας αυτό, έτσι, είναι καθημερινή υπόθεση. Όπως σας είπα είμαστε μια βιομηχανία που συνεχώς ανακυκλώνει τα πάντα, οτιδήποτε είναι υποπροϊόν μιας διαδικασίας ε, ξαναχρησιμοποιείται σε, άλλη, σε άλλο εργοστάσιο. Να σας δώσω τι να πω, από τη δεκαετία του 1880 ε, είχε ξεκινήσει αυτή η υπόθεση με... από όταν ξεκίνησε η χημική βιομηχανία. Λοιπόν, κύριε Τούρμες, θέσατε το ερώτημα τις τιμές χονδρικής και με τις πραγματικές τιμές το τι γίνεται. Δυστυχώς πρέπει να πω, και αυτό αφορά και την κυρία Νίμπλερ, Καμιά φορά, ε, τι να σου πω, δηλαδή μιλάνε οι τυφλοί για τα χρώματα. Έμα ε, τα κάνουμε όλα σαλάτα, δεν μπορώ και εγώ να σας απαντήσω σοβαρά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ως ε, άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζομαι εργοστάσια τα οποία δουλεύουν 24 ώρες, σε 24 ώρη βάση και μόνο έτσι μπορούν να αποδώσουν, δεν μπορώ να αγοράσω ρεύμα στην αγορά του σποτ ε, επειδή είναι φτηνότερο. Κάνω μακροπρόθεσμα συμβόλαια και δεν ε, καλύπτονται από αυτές τις καμπύλες τις οποίες ε, βλέπετε. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν σχέση τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε εσείς με την δική μας την κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να τα δείτε. Γι' αυτό ακριβώς συνέκρινα το επιχειρηματικό περιβάλλον σε ΙΠΑ και Γερμανία. Και αυτά ακριβώς τα είχα πει και στο Υπουργείο στο Βερολίνο. Αυτή τη σύγκριση που κάνουμε εμείς για να κρίνουμε πού θα φτιάξουμε ένα εργοστάσιο. Μετά για το ερώτημα του συνολικού κόστους της ενέργειας. Θα έλεγα συνολικά το κόστος ενέργειας είναι γύρω στο μεταξύ 21 και 22% ε, και αν βγάλουμε μάλιστα και την ε, παραγωγή των ε, βασικών υλών είμαστε στο 31%. Λοιπόν, για το προηγούμενο πάνελ πράγματι είπαμε ότι ανακατεύουμε κάποια διαφορετικά πράγματα και είπατε τι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω στην ενεργειακή αποδοτικότητα πράγμα το κάνουμε, αλλά πλέον ο ρυθμός της αύξησης, της αποδοτικότητας δεν θα είναι τόσο μεγάλος όσο ήταν στην ε, αρχή. Γιατί στην αρχή μπορούσαν να γίνουν οι μεγάλες ε, εξοικονομήσεις και θα έχουμε τώρα μία αύξηση ένα το πολύ 2% το χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί χρονικό πλαίσιο μιλάμε για να μιλήσουμε για μια σοβαρή εξοικονόμηση. Θα πρέπει να το δούμε αυτό σχέση και με τον κύκλο των ε, επενδύσεων. Δηλαδή όταν κάνουμε και μια επένδυση αντικατάστασης αυτό δεν γίνεται ε, σε ένα χρόνο ούτε, γίνεται, ε, ούτε γίνονται όλα μαζί. Μετά, τελευταία ερώτηση ήταν η τιμή του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτή τη στιγμή σήμερα έχουμε μια τιμή γύρω στα 8 ευρώ για το πιστοποιητικό. Έχουμε λοιπόν 200 εκατομμύρια κόστος στην ε, Γερμανία. Αν πάμε σε μία τιμή όπως θέλει η Κομισιόν μετά τη μεταρρύθμιση 40 ευρώ, αυτό σημαίνει θα πάμε στα 2,2 δισεκατομμύρια κόστος για την βιομηχανία. Βλέπετε λοιπόν το τεράστιο αντίκτυπο που σημαίνει το να ανέβει τιμή από τα 8 και 10 ευρώ στα 40. Δεν ε, απαντήσατε στην ερώτηση για τις διεθνείς, ε, τα διεθνή δικαιώματα εκπομπών. Ο κ. Μασιμιλιάνου Μασιμιλιάνο σας ε, πήδησα γιατί ήσασταν στο πίσω μέρος της σελίδα γραμμένο το όνομά σας. Δεν πειράζει, Πρόεδρε. Πολύ σύντομος θα είμαι και ευγενής. Δεν θέλω να είμαι προκλητικός γιατί με αντιμετώπισα μεγάλη ευγένεια και αυτό θέλω να το ανταποδώσω. Και δεν θέλω να είμαι προκλητικό. Δύο σχόλια τάχιστα. Πρώτον, το θέμα του ενεργειακού κόστου είναι μεγάλη απειλή, αλλά είναι η δεύτερη απειλή για την Ιταλική βιομηχανία. Όχι και Ευρωπαϊκή Διαφωνία Πρώτον, η πρώτη απειλή, κατά την άποψή μου, προέρχεται από του κινδύνους που συνδέονται με την αναγνώριση του καθεστώτος της οικονομίας της αγοράς της Κίνας. Επίσης, το ενεργειακό σύστημα αναμένοντας την πραγματική ενεργειακή ένωση, έχει διάφορα προβλήματα. Δύο. Το, το πρώτο το ανέφεραν πάρα πολλοί ομιλητές και αφορά το θέμα της ε, ενιαίας ε, τιμής που καταβάλουν τουλάχιστον οι ανεγροβόρες ε, επιχειρήσεις. Και δεύτερον, το, της αντιστάθμισης των έμεσων δαπανών. Εγώ είμαι επιβεβαισμένος ότι χρειάζεται να υπάρξει πραγματική αντιστάθμιση των δαπάνων αυτών. Γιατί ξέρουμε στην Ευρώπη ότι υπάρχουν ε, οι καλές και οι κακές χώρες. Βλέπω, είμαι περιστοιχισμένο από Γερμανού. Η Γερμανία είναι καλός μαθητής. Η δική μου χώρα, η Ιταλία, είναι κακός μαθητής. Δεν νομίζετε ότι στα πλαίσια τη αντισταθμίση ε, του αέμεσου κόστου μπορούμε να, με μεγαλύτερη ας πούμε, ε, εναρμόνιση, να διευκολύνουμε τις ενεργοβόρες ε, επιχειρήσεις. Ο κ. Σαμαδάρ. Ευχαριστώ. Πρώτο ερώτημα του κ. Νίκα. Έχω απλή απάντηση. Κανένα από τα δικά μας σχέδια στην εταιρεία δεν μπόρεσαν να σεβαστούν τα benchmark. Και κανένα στη Χαλιβουργία δεν μπορεί να σεβαστεί, δεν έχει το επίπεδο τεχνολογίας για να σεβαστεί τα, τα πρότυπα αυτά του ETS. Κάποια από αυτά τα εξήγησα στην παρέμβασή μου και αυτό βεβαίως πρέπει να διορθωθεί. Για το θέμα της ε, υπέρβασης των δικαιωμάτων εκπομπών, στις αρχαικές φάσεις του προγράμματος, NAT 1 και NAT 2, αυτή η υπέρβαση οφειλόταν στην τότε κρίση που είχαμε. Δεν θέλουμε να υπάρχει κρίση, γιατί επλήγει και η βιομηχανία και πολλές από τις επιχειρήσεις. Τα έσοδα που είχαμε από, τα, από τις υπερβάσεις επενδύθηκαν για ε, επενδύσεις ε, εντάσσεως ενέργειας, ούτως ώστε να ετοιμαστούν αυτές οι επιχειρήσεις για τους μηχανισμούς του ETS. Και συνεχεία η βιομηχανία και εμείς ξαναγοράζει δικαιώματα για να προχωρήσει τα προγράμματά της και δεν υπάρχει κανένα hedging, καμία αντιστάθμιση κινδύνου. Ε, μετά το 2020 μπορεί να μην έχουμε άλλα δικαιώματα και αυτό είναι πρόβλημα για μας. Για τις προτεραιότητες τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το μέγεθος και η ένταση του προβλήματος ε, δεν είναι στατικό. Αλλάζει, είναι δυναμικό. Η Κίνα και η αναγνώριση του καθεστώτος οικονομίας ε, της αγοράς είναι μεγάλο θέμα. Η παρουσίασή μου ανέφερε για ένα σενάριο που προβλέπουμε μετά το 2020. Γι' αυτό δεν σας είπα πολλά για την Κίνα. Ε, πάντως, με δεδομένη την κατάσταση, η Κίνα είναι από τα μεγάλα μας προβλήματα. θα γίνει με, τις, ε, με τη διαμόρφωση των τιμών. Ή μάλλον δεν είναι οι τιμές αυτές καθεαυτές, είναι αν θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε μέσα σε ένα δίκαιο πλαίσιο. Αν υπάρχει δικαιοσύνη, τότε το περιθώριο που έχουμε θα μας ε, δώσει τη δυνατότητα να επανεπενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες και να σεβαστούμε τη τα όσα μας λέει η Κομισιόν, ούτω ώστε να υποφεληθούμε από το ETS. Αλλά δεν έχουμε τέτοιο περιθώριο στον κλάδο μας. Είμαστε σε δύσκολη θέση και επιπλέον, εάν προσθέσουμε και την έλλειψη ισοτιμίας που υπάρχει, δηλαδή έχουμε χάλιβα που εισάγεται από άλλες χώρες στην Ευρώπη χωρίς να πληρώνουν ας πούμε, για τις εκπομπές ε, του διοξιδίου του άνθρακα που εμείς θα πληρώνουμε μέχρι το 2020, ε, αυτό μας ε, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή είναι η απάντησή μου, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. You're Τεγκέστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποσχέθηκα ότι θα απαντήσω όλα τα ερωτήματα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα για την ενεργειακή απόδοση. Η ενεργειακή απόδοση εξακολουθεί να είναι στο DNA της βιομηχανίας ε, του κλάδου μας και στην BASF, την εταιρεία μου. Δύο πράγματα να πω. Πρώτον, πρέπει να κάνουμε αυτά που μας αναλογούν και να ε, προσαρμόσουμε τα, ε, τις μονάδες μας, το ISO, το καινούριο πρότυπο και δεύτερον, χαίρομαι, θα εστιάσουμε περισσότερο στην ενεργειακή απόδοση και σε τομεί που δεν έχουν να κάνουν με το ETS. Και έτσι θα δείτε, αν εστιάσετε εκεί, που ε, και πόσο συμβάλλουν τα χημικά προϊόντα και η χημική βιομηχανία σε άλλους τομείς που εξακολουθούμε να μπορούμε να πετύχουμε πολλά με την ενεργειακή απόδοση, κατοικία, μεταφορές και πολλοί άλλοι τομείς. Άρα, ενεργειακή απόδοση είναι στο επίκεντρο του κλάδου. Δεύτερον, τιμή του δεξιδίου του άνθρακα. Φυσικά, εμείς χαιρόμαστε όταν θα έχουμε μια παγκόσμια τιμή για τις εκπομπές του άνθρακα, αλλά η λέξη κλειδί είναι παγκόσμιες. Ε, και είδαμε τι έγινε και στην COP21 στο Παρίσι για πρώτη φορά επιτεύχθη μια παγκόσμια συμφωνία. Να την εφαρμόσουμε πρώτα όμω αυτή την παγκόσμια συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά χωρί να χάσουμε την ανταγωνιστικότητα ε, στην Ευρώπη και βέβαια στην κυκλική οικονομία. Δεν έχουμε μόνο αυτή την έννοια fair bund, αλλά έχουμε και τα, ανακάνουμε με τα προϊόντα τα οποία αναπτύσσουμε. Όταν βλέπουμε ότι το 1 τρίτο του προπολογισμού ενό ομίλου όπω η BASF πηγαίνει εκεί, σε αυτή την κατεύθυνση, εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένο ότι η κυκλική οικονομία θα είναι ένα παράγον κλειδί για την επιτυχία όλων των βιομηχανιών από κοινού, αλλά βέβαια θα πρέπει να δούμε και την αλυσίδα της αξίας, όχι ενό κλάδου όλων των κλάδων της βιομηχανίας. Υποσχέθηκα να είμαι σύντομος κύριος Τούρμης. Να μας δείξετε λένε. ναι. Ευχαριστώ τον κύριο Ντε Θα δώσω το λόγο για μια ακόμη φορά στον κύριο Τίλμαν, αλλά προηγουμένως να σας θυμίσω αγαπητοί συνάδελφοι ότι είχαμε εκπροσώπους της ε, επιστημονικής κοινότητας και στα δύο μέρη του πάνελ. Είχαμε τον καθηγητή Νόηχο στο πρώτο πάνελ και τον δόκτωρα Τίλμαν στο δεύτερο. που έχει μεταδιδακτορική θέση στο Ινστιτούτο. Έχει κάνει επιστημονική δουλειά στο Πολυτεχνείο. Ε, μπορείτε αυτά να τα βρείτε στο βιογραφικό του και να τα μελετήσετε πολύ προσεκτικά. Άρα υπήρξε απόλυτη ισορροπία στα μέλη του πάνελ και των δύο πάνελ. Εγώ δεν λέω αερολογίες, μιλάω με στοιχεία. Τώρα, ε, μπορείτε να απαντήσω ο κ. Σάλιν, κύριε Τίλμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ρωτήσατε το τι γίνεται με την ε, αποζημίωση αυτή την αντιστάθμιση. Εμείς λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή στη Γερμανία 160 εκατομμύρια όσον αφορά τα πιστοποιητικά, το έμεσο κόστος. Και βεβαίως βλέπουμε στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας πως ε, ε, θα έπρεπε να το κάνουν και άλλες χώρες. Το θέμα είναι όμως ότι μέχρι σήμερα δεν είναι ξεκάθαρο το τι θα γίνει από εδώ και προς. γιατί προσεχώς αν πάει στα 2,2 δισεκατομμύρια θα φτάσουμε, θα εμείς θα έχουμε μόνο 600 εκατομμύρια αντιστάθμιση οπότε βλέπετε πως αφενός τώρα παίρνουμε κάτι αλλά στο μέλλον θα λαμβάνουμε πολύ λιγότερο και βέβαια έχετε δίκιο πρέπει να ισχύσει για όλους Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ πάρα πολύ Ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη του πάνελ και πηγαίνουμε στις καταληκτικές παρατηρήσεις που θα μας κάνει ο κύριος ε, Ντομινίκ Ριστόρη, γάμα δέλτα, της, ε, γενικός διευθύνσης γάμα δέλτα, ε, ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΙΤΡΕ. Το ενεργειακό κόστος και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας είναι σημαντικές προκλήσεις. Νομίζω όμως ότι είναι καλό να πάρουμε κάποια απόσταση από κάποια επίμαχα ζητήματα και να εξετάσουμε τι έχουμε πετύχει στην Ευρώπη. Χάρη στην ευρωπαϊκή πολιτική εν γέννη, αλλά και ειδικότερα χάρη στην ενεργειακή ευρωπαϊκή πολιτική. Πρώτα απ' όλα, κατέστη δυνατόν να εξασφαλίσουμε την αποσύνδεση το διαχωρισμό της οικονομικής ανάπτυξης από την κατανάλωση της ενέργειας. Αποσυνδέσαμε, διαχωρίσαμε αυτά τα δύο πηγαίνοντας στην κατεύθυνση. And let me say, uh, certainly, European Union industry has used της ενεργειακής απόδοσης. Η πιο... Our main competitors. This is crystal clear. Εμείς είμαστε πιο αποτελεσματικοί στη χρήση της ενέργειας. Ε, αυτό προκύπτει από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων που έχουμε για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις εδώ και 20 χρόνια. Η εντύπωσή μου είναι ότι οι νέες τεχνολογίες, κυρίως το χάλιβας, ε, κατασκευαστικός τομέας, χημική βιομηχανία, έχουν πραγματικό δυναμικό να βελτιώσουν περαιτέρω την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και θα πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Γιατί πραγματικά κάνει τη διαφορά. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Τα τελευταία δύο χρόνια μειώσαμε το χάσμα ανάμεσα στις τιμές χοντρικής με τους βασικούς μας ανταγωνιστές, κυρίως Αμερικανούς. Αυτό προκύπτει αν εξετάσουμε την κατάσταση των τιμών ε, χονδρικής ενέργειας είναι το 1,7 της τιμής χονδρικής της, Αμερι... Ε, της αμερικανικής αγοράς. Ενώ το 2013 είμαστε στο 2,5% ή στο 3%. Ε, συγγνώμη, στο 2, ήταν 2,5 φορές παραπάνω ή 3 φορές παραπάνω. Και το ίδιο για τις τιμές χονδρικής του φυσικού αερίου παρότι το χάσμα ανάμεσα μας και τους Αμερικανούς εξακολουθεί να είναι μεγάλο. Τρίτη παρατήρηση. Σημαντικό να δούμε τις διαφορετικές συνιστώσεις των τιμών ενέργειας. Γιατί είναι αλήθεια ότι αν για πολλές τιμές λιανικής της ενέργειας. Είμαστε στο 40% των μη ενεργειακών δαπανών. Είναι σημαντικό να ανοίξουμε τη συζήτηση εδώ στα κράτη-μέλη και να συζητήσουν όχι μόνο οι Υπουργοί Ενέργειας, αλλά όλοι Λίβαν. As you know, we have decided to... Αποφασίσαμε, όπως ξέρουμε, να κάνουμε μια βαθιά ανάλυση των ε, τιμών ενέργειας και του κόστους ενέργειας. Η πρώτη μελέτη παρουσιάστηκε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και θα επικαιροποιήσουμε αυτή την ανάλυση και θα παρουσιάσουμε το καλοκαίρι τα τελικά αποτελέσματα. είναι σημαντικό να τα συζητήσουμε όλα αυτά και στο Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο. Και να θυμίσουμε στα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν τις πραγματικές ε, ενεργειακές τιμές και δαπάνες στη λεγόμενη ενεργειακή διακυβέρνηση, στο Energy Governance. Και θα γίνει αυτό το πράγμα, θα αποτελέσει ένα σημαντικό δίκτυο για την ενέργεια. Ξέρω, ότι εσείς Πρόεδρε και η Επιτροπή σας σε ό,τι αφορά το Energy Governance θέλετε να δείτε τις προτάσεις που θα παρουσιάσουμε μέσα στο 2016. Και θα πρέπει να γίνει μια σημαντική συζήτηση για να διαπραγματευτούμε το ενεργειακό και κλιματικό πλαίσιο για το 2030 στα πλαίσια του Συμβουλίου του Οκτωβρίου. Τώρα πρέπει να το ενσωματώσουμε το στοιχείο ως, γιατί είναι βασικός δείκτης. Τέταρτη παρατήρηση. Οι νέες προτάσεις που θα παρουσιάσουμε μέσα στο 2016 θα συνεισφέρουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ενεργειακού κλάδου. Όπως ξέρετε, θα παρουσιάσουμε το νέο σχεδιασμό της αγοράς. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα μιλήσουμε για αυτή την έννοια και θα συμφιλιώσουμε την αυξανόμενη, το αυξανόμενο μερίδιο των ανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά και ταυτόχρονα θα εξασφαλίσουμε τις επενδύσεις, τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα για τους καταναλωτές. Θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο δραστήρια στο νέο ενεργειακό πανόραμα. Αυτή θα είναι μια πραγματική ενεργειακή επανάσταση, γιατί ξέρετε ότι από την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού οι καταναλωτές πληρώνουν τον λογαριασμό, regarding the energy consumption, including the time of consumption. And this will be important. Τώρα, εμείς θα επιλέξουμε την καταναλώσή μας. Και αυτό είναι σημαντικό για την ατομική και συλλογική κερδοφορία του κλάδου, του ενεργειακού κλάδου. Επίσης θα προτείνουμε να εξασφαλίσουμε περαιτέρω ε, ενεργειακή αποδοτικότητα μέσω της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα και θα κάνουμε και διάφορα πράγματα για να διευκολύνουμε τις επενδύσεις γιατί έχουμε πολλά καλά project για την ενεργειακή αποδοτικότητα, για τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, αλλά και για τη διαλειτουργικότητα των υποδομών ηλεκτρισμού και ψυχού αερίου. Και πρέπει να κατασκευάσουμε, να χτίσουμε αυτή τη νέα γέφυρα ανάμεσα στους, σε αυτούς που προωθούν αυτά τα προγράμματα και στους επενδυτές. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι η βασική συνεισφορά. Όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αλλά και των εθνικών τραπεζών και, ε, τραπεζών και όλων των ε, εθνικών φορέων για να αναπτύξουμε και να προωθήσουμε την ε, συνολική μας ανταγωνιστικότητα. Και είμαι πεπισμένος ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα νέο επίπεδο ισότιμου ανταγωνισμού και να τελειώσουμε κάτι θετικό. Ο συνάδελφος βρίσκεται στην Αμβέρσα. Στην Αμβέρσα έχουμε μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία που αποφάσισε να επενδύσει στον τομέα των δηληστηρίων. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Τώρα το αποφάσισε. Τώρα, μόλις, θετικό το μήνυμα ό,τι αφορά την ε, οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος αυτού. Δεν φαντάζομαι ότι αυτή η εταιρεία πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς να σκεφτεί το οικονομικό της όφελος. Και αυτό είναι θετικό μήμα. Και αυτό μας δίνει ακόμα περισσότερα κίνητρα για να προχωρήσουμε, για να έχουμε ένα στεναρό, σταθερό νομικό πλαίσιο, ούτω ώστε να προωθήσουμε ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά μας και να μειώσουμε ακόμα περισσότερο το κόστος της ενέργειας. Uh, thank you, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γενικέ Διευθυντά και για τις ε, παρατηρήσεις σας. Νομίζω πως ήταν πάρα πολύ σημαντικές, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ακρόαση. Σας ευχαριστώ όλους ε, και βεβαίως πρώτα απ' όλα τα μέλη του πάνελ, τους ομιλητές μας όλους σας. Άλλοι δύο ε, είναι στην αίθουσα. Πέντε συνολικά. Πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγισή σας ε, και το μήνυμα σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ε, παρακαλώ χειροκροτήστε. Thank And, uh, uh, uh, it is Λοιπόν, λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής. Έχετε να πείτε τίποτα άλλο. Στα διάφορα, όχι. Επόμενη συνεδρίαση 16-17 Μαρτίου. Πω πω Παναγία μου, μεγάλο διάλειμμα. Τρεις εβδομάδες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, διαλυθείτε ησύχως. Τώρα, για να ξεκινήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Κάποιοι θα μείνουν λοιπόν.